ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τα θύματα του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Ιαπωνία την προηγούμενη Παρασκευή και για τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αστέγους. Ενός λεπτού σιγή παρακαλώ. Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω ότι προτίθεμαι να αποστείλω μία επιστολή εξ ονόματός σας στο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας για να τους συμπαρασταθούμε στη δύσκολη αυτή στιγμή που διανύουν. Το Προεδρείο της ΑΦΕΤ αποφάσισε σχετικά με το πρωτόκολλο για την Ουκρανία στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο αυτό θα εγκριθεί με την απλουστευμένη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού χωρίς τροπολογίες. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορώ να θεωρήσω ότι έχει εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο και το θέμα θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου, τη Συνόδου του Απριλίου. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα θεωρούμε το θέμα αυτό ως λήξαν. Μου ανακοινώθηκε μου κοινοποιήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή στις ψηφοφορίες, διότι όσον αφορά την έκθεση David υπάρχουν ομάδες που θα πρέπει να ετοιμάσουν την, τον κατάλογο ψηφοφοριών. Γι' αυτό θα περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Σίβιτς πριν από την έκθεση Δαβίδ η οποία θα έχει και τον κατάλογο ψηφοφοριών των φιλελευθέρων που δεν υπήρχε μέχρι τούδε. Λοιπόν, βάλτε τις κάρτες σας και μπορούμε να αρχίσουμε. Ο κύριος Σίβιτς ε, ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνοψίσω την, ε, τις εργασίες μας και που θα ολοκληρωθούν σήμερα με τη σημερινή ψηφοφορία. Δεν έχουμε φυσικά χρόνο για συζήτηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν θέματα προς συζήτηση. Επιτρέψτε μου λοιπόν μόνο κάποιες λέξεις. Διάφορες ε, φορές συναντήθηκα με τους κοιόδες εισηγητές και οι διαπραγματεύσεις μας ήταν πάρα πολύ εντατικές οι τροπολογίες ξεπέρασαν τους 200 στον αριθμό, αλλά χάρη στην καλή θέληση και στη σκληρή δουλειά καταφέραμε να περιορίσουμε τον αριθμό αυτό με πάρα πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Υπήρξε καλό πνεύμα συνεργασίας κατά τις συναντήσεις αυτές. Και σε πολλές περιπτώσεις οι σκιώδεις εισηγητές εκπροσωπήθηκαν από εμπειρογνώμονες το οποίο και διευκόλυνε τις εργασίες μας με μία συγκεκριμένη εξαίρεση, την οποία αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε. Έχουμε την κυρία Τζόκοου, η οποία εκπροσωπεί το ΕΕΛΚ. Να την ευχαριστήσω προσωπικά για την παρουσία της κατά τη διάρκεια όλων των συναντήσεων μέχρι χτες το μεσημέρι. Είχαμε μία εκδοχή του κειμένου έτοιμοι για ψήφιση με ένα πολύ σαφές μήνυμα και είμαστε ενωμένοι μεταξύ των μεγάλων ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι υποστηρίζαμε την έκθεση. Ωστόσο, το απόγευμα το ΕΛΚ ε, την υποστήριξή του για δύο συμβαστικές τροπολογίες. Και οι δύο τροπολογίες αυτές είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι διταράχτηκε η ισορροπία. Όπως ξέρετε, ο συμβιβασμό ε, έχει να κάνει και με την υποχώρηση. Όταν αποσύρεται κανείς και δεν υποστηρίζει πλέον μια σεμιβαστική τροπολογία αργά το απόγευμα και τελικά δεν έχει κανείς χρόνο να βρει κάτι άλλο συμβαστική λύση, ε, να πω, είναι πολύ ατυχές αυτό. Δεν ανταποκρίνεται στην πολιτική κουλτούρα στην οποία έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι μας εκβίασαν κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό λοιπόν σήμερα όταν θα ψηφίσουμε θα είναι κατακαιρματισμένοι η ψηφοφορία αναφορικά με τους συμβιβασμούς και αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, απόσυρσης ε, του ΕΛΚ από, τους, ε, από τις συμβαστικές. Παρουσιάσαμε τα επιχειρήματά μας, αλλά οι, οι εταίροι μας από το ΕΛΚ κόφευσαν. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια αντίδραση, Τι να πω, θα πρέπει να αποφασίσουμε στην ψηφοφορία εν τέλει. Δεν προβλέπεται συζήτηση επί του θέματος. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπρόκ, ο οποίος θα μιλήσει εξ ονόματος της ομάδος και κλείνει η συζήτηση. Κύριε Μπρόκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ το ότι δεν είναι ικανοποιημένο ο κύριος Σίβιτ για το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές αποκλίνουσες απόψεις αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά απόλυτα φυσιολογικό όταν έχουν κατατεθεί συμβαστικές προτάσεις να συζητηθούν από τις πολιτικές ομάδες. Και σε τέτοια περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτά τα πάντα, αλλά Ορισμένοι εκφράζουν επιθυμίες για τροποποίησης. Νομίζω ότι με κάποια καλή θέληση μπορούμε να καταλήξουμε σε μια μέση οδό και έτσι σε ένα αποτέλεσμα. Λυπούμε για τις αντιδράσεις του κυρίου Σίβιτς. Εμείς διαθέτουμε την βούληση να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να λησμονούμε και την δημοκρατία εντός της πολιτικής μα ομάδας. Και είμαι βέβαιο ότι η κυρία Γιαννάκου έκανε σημαντική προσπάθεια. Σε δύο σημεία έχει μια κάπως διαφορετική τοποθέτηση. Δεν θα πρέπει τώρα να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις και να ομιλούν εδώ ορισμένοι για την πολιτική των ισχυρών και άλλα τέτοια. Μίλησε ο εισηγητής και η ομάδα. Να μου πείτε σε ποιο άρθρο βασίζεστε και πού θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό ζήτημα για αυτή τη μικρή αλλαγή ως προς τις πληροφορίες. Δεν ήταν όλα ορθά που ακούσαμε. Αυτή η απόσυρση του ΕΛΚ από την παράγραφο 5 και από τις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες δεν ήταν απόφαση της ομάδας, δεν ψηφίστηκε ποτέ στην ομάδα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, νίκη της δημοκρατίας. E- λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Θα δούμε πώς έχει η δημοκρατία και πώς ορίζεται γιατί θα ψηφίσετε. Όχι καμία συζήτηση, καμία συζήτηση. Παράγραφος 1, τροπολογία 36. Παρακαλώ, υπέρ. Διανατάσεως, υπέρ. 36, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ παρακαλώ κατά δεν είναι σαφές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 41 αρχίζει η ψηφοφορία Chiusa la votazione. Πέρας υπέρ 23, κατά 33, απορρίπτεται 42. Αποσύρεται 43 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 44, αποσύρεται 45 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Ανοίγει η ψηφοφορία επί της 49. Chiusa la votazione. Peras. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Votazione. Si adottato. Ah no, Eh, Κλείνουμε, λείπουν τρεις ψήφοι. 30-26 απορρισσύρεται 52, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2 στην 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Υπέρ της 60. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι απόλυτα σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 63. Chiusa la votazione. Πέρας. Υπέρ 27, 34 κατά απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 Α, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος 69 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 70. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80, 80 τώρα υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, επί της 80. Πέρας. 36 κατά. Απορρίπτεται. Voti contrari.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 νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική κλίση, ονομαστική κλίση. Επί της 94 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία πάλι. Είχα ορισμένες αμφιβολίες. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά. Και εδώ δεν είναι απόλυτα σαφές. Θα πρέπει να ελέγξουμε, αρχίζει η ψηφοφορία για την 95. Πέρας. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επί της 102, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Υπέρ της 3, κατά, αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4. Α, θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 114. Πέρας. Πέρας. 38 ναι, όχι 24. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 126. Πέρας. Αυτή φορά ψήφισαν όλοι. Για μία ψήφο απορρίφθηκε. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 133 Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 138. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 144 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ε, απορρίφθηκε 146 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 148 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 149 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 151 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 153 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 154 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 157. Όχι, όχι, όχι, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε για 154. Άρα πάμε στην 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 159. Προφορική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα της 160. Chiusa la Πέρας. Εγκρίνεται. 37 έναντι 24. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 165 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ψηφίσουμε 182 με ονομαστική κλίση πέρας ε, ε, ε, ισοψηφία ισοψηφία Άρα απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγώ λέω εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Θέλετε να ελέγξουμε, ευχαρίστως. 188 με ονομαστική κλίση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αν το επιθυμείτε, βεβαίως. Πέρας. 45 υπέρ. Θα αλλάξω γυαλιά, λέει ο πρόεδρος. 45-19. 188 λέει υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 189 λέει ο πρόεδρος. 189 γιατί την 188 την ψηφίσαμε με ηλεκτρονική. Quasi tutti, eccetto ecco adesso ha votato anche l'uno, 44 no. Απορρίπτεται. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται η 11 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά δεν είναι σαφές 19 αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας Πράγματι απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 22. Chiusa Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 31 υπέρ. Κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος. Για άλλη μια φορά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε επί της 31. Όλοι ψηφίσανε 32 έναντι 31. Εγκρίνεται για μια ψήφο. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1. Α, θέλετε να ελέγξουμε τη 35, εντάξει, αρχίζει η ψηφοφορία επί της 35.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 Πέρας. Εγκρίνεται 61 υπέρ, 1 κατά. Δύο αποχές. Να συγχαρούμε λοιπόν τον εισηγητή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης David. Στο μεταξύ έχουμε και τον κατάλογο ψηφοφοριών ακόμα και για τις ε, ομάδες έννοιες που δεν είχαν τον κατάλογο, μπορούμε να αρχίσουμε με την ψηφοφορία αν επικρατήσει λίγη ησυχία. Ο κύριος Βιγγένιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό μόνο. Ε, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σας ζητήσω στο μέλλον όταν, όταν έχουμε οι συνεδριάσεις ε, της Επιτροπή μα, να μην ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες γιατί είδατε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα. Τελευταία στιγμή δεν είχαμε χρόνο στη διάθεσή μα να συζητήσουμε και τα θέματα περί ανατολικής ε, πολιτικής. Κάποιες ομάδες δεν είχαν τον κατάλογο ψηφοφορίας για το Νότο, να σας παρακαλέσω να βάζουμε τις ψηφοφορίες το απόγευμα. Και κατά δεύτερον, είχαμε την αίσθηση ότι καλή ιδέα θα ήταν να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Ολομόλια, να μην ψηφιστεί στο Στρασβούργο, αλλά στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. αυτό για να σας αναφέρω ποια είναι η άποψη των σοσιαλιστών και δημοκρατών στην Επιτροπή μας, για να έχουμε πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δηλαδή να συζητήσουμε την έκθεση. Ως προς τη δεύτερη αντίρρηση, η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει επί του χρονοδιαγράμματος. Ως προς την πρώτη αντίρρηση, αντίρρησή σας θα μπορούσε να γίνει το απόγευμα, αλλά επειδή είχαμε άλλες ακροάσεις, υπουργού και ούτω καθεξής, έπρεπε να λάβουμε υπόψη αυτούς τους ε, περιορισμούς χρόνου. Αλλά όταν δεν υπάρχουν τέτοια θέματα θα το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να ε, ψηφίσουμε κύριε Σίβιτς, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. 30 δευτερόλεπτα. Αυστηρά. Μόνο 15 δευτερόλεπτα θα χρειαστώ. Υποστηρίζω την ιδέα να αναβληθεί η ψηφοφορία στο Στρασβούργο, γιατί θα μα δώσει ευκαιρία να συνάψουμε μεγαλύτερου συμβιβασμού. Και αν συμφωνήσει και ο κύριο Ντάβιτ, ζητούμε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Να μην γίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά στο Στρασβούργο. Ε, Συμβιβασμό 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται 61, 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 ήταν σαφές αν θέλετε ελέγχουμε την 64 αρχίζει η ψηφοφορία Ψηφίζουμε την 64 για την 64. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. 36 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αποσύρεται. 68 υπέρ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 Θέλετε να ελέγξουμε την 72. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. 32 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75. Α, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 αποσύρεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100 με την προφορική γκόμες υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται 101, 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 106 με την προφορική κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Άρα ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση επί της 110. Λείπουν τρεις ψήφοι, αλλά κλείνουμε. Εγκρίνεται. 33 υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται, 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113. Α, όχι, όχι. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Θέλεις να παρέμβεις ο κύριος Νταβίτ. Να ρωτήσω τους συναδέλφους κατά πόσο θα μπορούσαν να αποδεχτούν μια προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας αυτής. Την εξής ανησυχεί για το status quo σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσογείου και ζητά διαπραγματεύσεις. Αυτές τις ε, λέξεις προσθέτουμε όταν οι όροι πληρούνται για ε, μια βαθιά ζώνη ε, ελεύθερου εμπορίου. Να προσθέσουμε δηλαδή το when requirements are met, όταν πληρούνται οι όροι. Eh, Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να ψηφίσουμε με αυτή την προστίκη. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ωραία, ελέγχουμε αν το επιθυμείτε. 137. Ελέγχουμε.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 αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται 167-168 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται 170-171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 178 όχι, με συγχωρείτε, κάνω λάθος. Συμβιβασμός 11 λέει ο πρόεδρος, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 υπέρ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 κατά, αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 39 με την προφορική του εισηγητή υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 40 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 41 υπέρ Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την 40. Αρχίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία από τη 40.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 αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 α όχι όχι καταπίπτει γιατί δεχτήκαμε τη 13 άρα προφορική 0α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 16 υπέρ Α, κάτι θέλει να μας πει ο εισηγητής πριν ψηφίσουμε την 16 Πρόεδρε, να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος. 11 ε, Μαρτίου είναι η ημερομηνία για το ψήφισμα για τη Λιβύη, όχι 10 Μαρτίου. Ε, εντάξει, θα καταγραφεί. Ψηφίζουμε επί του συμβασμού 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 4, 4, 5 και 6 μαζί, το δέχεστε εντάξει, 4, 5 και 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, αποσύρεται 7, καταπίπτει η 8, ψηφίζουμε την 9, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου της έκθεσης David. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν, αν και δεν έχουν ψηφίσει δύο, 58 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές, συγχαρητήρια στον κύριο Νταβίντ. Για το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα, στο επόμενο σημείο της, κυρία, της ε, ημερήσιας διάταξης έχουμε την ακρόασή μας, ο κύριος Νέης. Κυρία. Η κυρία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, επιτρέψτε μου πρώτα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντάβιντ για την μόλις εγκριθήσα έκθεσή του. Ωστόσο, θα προτιμούσαμε να αναβληθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια μέχρι την περίοδο συνόδου του Στρασβούργου, ώστε να προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα κείμενα στην ταχεία εξέλιξη των γεγονότων. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα καταψηφίσουμε, γιατί ψηφίσαμε υπέρ τη εκθέσεω. Ωραία. Το καταγράφουμε. Ο κύριος Χάουιτ ζητάει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Χάουιτ. Εντάχει, εγώ ήμουν σκιώδης επί της ε, έκθεσης για τη συνεργασία στον ε, Περσικό κόλπο. Αν αφήσουμε το κείμενο ως έχει, τότε φαινόμαστε κάπως απαρχαιωμένοι. Ε, θα αποφασίσουν οι ομάδες αν θα αναβάλουμε ή όχι, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να αποφανθεί για ορισμένες προτάσεις συμβιβασμών στην Ολομέλεια έτσι ώστε να είμαστε επικαιροποιημένοι κάπως. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα ο συνάδελφος Άσκου να με αντικαταστήσει και του αναθέτω την Προεδρία. I'm stepping in. Okay. The, the beautiful, the beautiful President Castro. Hi. Buongiorno. How long do you want to speak? Because we are a bit...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 Okay, let's start because... αρχίσουμε, γιατί έχουμε ήδη μια καθυστέρηση 20 λεπτών. Είναι αρκετά φορτωμένη η ημερήσια διάταξή μας σήμερα και πρέπει να, την, να προλάβουμε να την εξαντλήσουμε. Θα ήθελα τώρα να απευθύνω το καλώς ορίσατε τον κύριο Βασκονόσκη που είναι αναπληρωτής υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, καλώ ήλθατε κύριε Υπουργέ. καθώ επίση απευθύνω το ορίσατε και στον κύριο Χάτζη Μαρκάκη που είναι ο πρόεδρο τη αντιπροσωπείας για τι σχέσει με την χώρα που εκπροσωπείται σήμερα εδώ κοντά μα. και καθώς επίσης και ε, τα υπόλοιπα μέλη της ε, αντιπροσωπείας αυτής. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι ο χρόνος είναι όριμος ε, να συζητηθεί η κατάσταση στην χώρα σας καθώς και η πρόοδος της υποψηφιότητάς σας και κατόπιν ως γνωρίζετε θα, συζητήσουμε, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την έκθεση πρόοδου για την χώρα σας. Ελπίζω στο τέλος της συζητήσεως αυτής όλοι να κατανοούμε καλύτερα την κατάσταση και να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε περαιτέρω. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προβείτε σε μια εισαγωγική ομιλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι σημαντική ευκαιρία αυτή για μας να μπορέσουμε να σας απευθύνουμε το λόγο σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσουμε τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις του 2010 στην Μακεδονία καθώς και το σχέδιο πρόοδου, εκθέσεως πρόοδου δηλαδή του κ. Ζόραν Τάλερ. Ευχαριστούμε πολύ ε, τον κύριο Τάλερ για την συμβολή του στην ευρωπαϊκή ατζέντα και στην ένταξη της χώρας μας. Είχαμε στενή συνεργασία με τον κύριο Τάλερ και αυτή θα συνεχιστεί και ε, στους επόμενους μήνες και ε, γενικά στην επόμενη περίοδο. Ορισμένες από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην χώρα μας θεωρούμε πολύ σημαντικό τον διάλογο που διεξάγουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωβουλευτές. Ορισμένοι έξι μόνο έχουν ήδη επισκεφθεί την χώρα μας. Συνεχίζουν να ε, συμβάλλουν σε μια μεγαλύτερη ε, γνώση και ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής μας ατζέντα και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε ανοιχτά και επικοδομητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ε, οι απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικές για μας και λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη από την από την ε, κυβέρνηση της ε, Μακεδονίας. 20 χρόνια πέρασαν από την ειρηνική απόσχηση της χώρας μας από την Ιουγκοσλαβία, η, η μόνη χώρα που ε, είχε την τύχη αυτή. Στα τελευταία 20 χρόνια η Μακεδονία απέδειξε ότι είναι αξιόπιστο σύμμαχος και πραγματικό σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε βρέθηκε, τάχθηκε με την σωστή πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κρίση της δεκαετίας του 90 στα Βαλκάνια και του 1999 στο Κόσοβο αλλά και σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής η χώρα μας πάντοτε τήρησε τις ίδιες ακριβώς θέσεις όπως η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ξεπεράσει κανένα από τα θεσμικά στάδια. Ξεκινήσαμε το 1996 από την Συμφωνία Συνδέσεως, μετά Συμφωνία Σταθερότητας ε, κατόπιν και μετά λάβαμε το 2005 το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας και το 2009 έγινε η σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμο ορόσημο. Αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη, δηλαδή πρόκειται να αρχίσουν. Η ευθύνη είναι δική μας να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την σημαντική ευκαιρία των υπολείπων θεσμών μας και των άλλων πολιτικών φορέων, αλλά είναι και μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Τα Βαλκάνια δεν είναι ούτε τμήμα της Αφρικής ούτε της Ασίας. Είναι τμήμα της Ευρώπης. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ρόλο και να αναλάβει τις ευθύνες της για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε αυτή την περιοχή. Η κυβέρνησή μας αποδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στην ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας μας που αποτελεί στρατηγικό στόχο όλων των κυβερνήσεών μας από την εποχή της ανεξαρτησίας μας. Υποστηρίζεται και από τους πολίτες, από όλες τις πολιτικές ελίτ, από τις μη κρατικές οργανώσεις, από τα μίντια και από όλους τους φορείς της κοινωνίας. Πιστεύω ότι η, σημερινή πλειοψηφία που εκπροσωπείται σήμερα είναι σημαντική, είναι αναγκαιότητα για την χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει και πολιτικά και οικονομικά πολύ σημαντικά στην περιοχή, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξεπηδήσουν νέοι κίνδυνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς που διαθέτει για να επιτρέψει τη χώρα να παραμείνει σε μια πορεία εντάξεως. Οποιαδήποτε αναστολή της διαδικασίας θα έχει αποθαρρυντικό αποτέλεσμα και κυρίως για τους νέους της χώρας μας οι οποίοι επιθυμούν να δουν την χώρα τους ως σύγχρονη χώρα να εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της ανοίγονται και ούτω καθεξής. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή των Βαλκανίων είναι μια ενεργός πολιτική διευρύνσεω που να βασίζεται στα προσόντα τη κάθε μια υποψήφια χώρας. Μπήκαμε με ενθουσιασμό στην συζήτηση για την πολιτική διεύρυνση. Μπήκαν βέβαια και διμερεί θέματα και έχουν οδηγήσει τώρα σε μια ανακοπή των προσπαθειών. Πρέπει να ξεπεραστούν τα πράγματα που μας διαιρούν, είτε γεωγραφικά είτε ιστορικά. Πρέπει να λυθούν ισότιμα και μέσα σε πνεύμα ευρωπαϊκής συνεργασίας όλα τα θέματα. Αυτά τα διμερεί θέματα στην ουσία κρατούν σιωμηρία την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές της, την πολιτική της διευρύνσεως που έχει προσφέρει τεράστια πλονεκτήματα σε εκατομμύρια πολιτών άλλων χωρών. Η προοπτική εντάξεως είναι ο ε, το πιο σημαντικό κίνητρο για την ε, πορεία προς με, τις απαραίτητες Είναι κρίσιμο, για την, είναι κρίσιμο η πορεία αυτή και για την σταθερότητα της περιοχής μας και για το μέλλον των χωρών μας. Αυτή η προοπτική πρέπει να παραμείνει προφανής, ορατή χρειάζεται και από τις δύο πλευρές τήρηση των υπεσχημένων και από την πλευρά την Ευρωπαϊκή και από την πλευρά των ε, ε, υποσχεδιών χωρών. Η Ουγγρική Προεδρία έχει τη σημαντική ευκαιρία να προωθήσει τα θέματα αυτά και άλλων βαλκανικών χωρών το ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Μακεδονία θα είναι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Έχουμε εργαστεί σκληρά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων εκπληρώντας τα απαραίτητα κριτήρια τα οποία όπως έχει αναγνωριστεί δύο χρόνια συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που τα συνέδεσε με την σύσταση να ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Όμως μπλοκαριζόμαστε λόγω της διαφωνίας για την ονομασία. διμερή ε, διμερές θέμα το οποίο ξεκίνησε από τη στάση μιας ε, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχουμε κάνει προσπάθειες με τους Έλληνες γείτονες να προχωρήσουμε και υπό την αιγίδα των Ενωμένων Εθνών. Η διμερείς ε, αυτή η διαφορά, ωστόσο δηλητηριάζει τις προσπάθειές μας. Προχωρούμε πάντως και με συνομιλίες υπό την αιγύδα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε άλλα πλαίσια με την συνεργασία των φίλων μας στην Ελλάδα για να βρεθεί μια διαρκής λύση που να είναι αποδεκτή και ε, από τις δύο χώρες και από τους λαούς των δύο χωρών. Μια λύση η οποία δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια οποιασδήποτε από τις δύο χώρες. Η ευρωπαϊκή ένταξη είναι η σημαντικότερη δύναμη που συγκρατεί και συνενώνει την πολυσχηδή κοινωνία μας. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή ε, πορεία ένταξης. Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό υπέρ της εντάξεως. Δεν ζητούμε ούτε shortcut ούτε fast track, ούτε δηλαδή να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια με ταχύ τρόπο θα πρέπει να διατηρηθεί το θετικό κλίμα στις μακεδονοελληνικές σχέσεις για να λυθεί η διμερής διαφορά με μια λύση διαρκή που να είναι αποδεκτή και από τις δύο χώρες και από τους δύο λαούς προς το συμφέρον της περιφέρειας αλλά και της ευρωπαϊκής σταθερότητας και ευημερίας. Ζητούμε και την υποστήριξη της Ελλάδος που είναι και το παλαιότερο κράτος μέλος στην περιοχή των Βαλκανίων με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης αλλά και με τη νέα πρωτοβουλία της Ατζέντα 2014. Ελπίζουμε η χώρα αυτή μέλος να δράσει υπεύθυνα και να χρησιμοποιήσει το δυναμικό της για να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της ε, ενταξιακής πορείας της περιοχής στην οποία ανήκει. Η Μακεδονία είναι ένα παράδειγμα της επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μεταξύ των υποψήφιων χωρών με καθαρή πολιτική βούληση, με καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες και σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις. Η Συμφωνία Σταθερότητας και σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμοστεί ομαλά. Μέχρι τον Ιανουάριο, 2000, τον Ιανουάριο 2011 προχωρήσαμε στην επόμενη συμφωνία και για το 2014 προβλέπουμε το επόμενο βήμα. Εμείς είμαστε, συμβάλλουμε και στην ασφάλεια στο International Crisis Management με 4% των δυνάμεών μας. Το 2011 είναι και ένα ορόσημο για άλλη σημαντική επέτειο της Μακεδονίας. Είναι η δέκατη επέτειος από τη Συμφωνία Πλαίσιο της Οχρίδας, αλλά και 15 χρόνια από την εξέλιξη των σχέσεων Μακεδονίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, έτος, το φετινό έτος θα πρέπει να θεωρηθεί κρίσιμο ορόσημο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να έρθω σε δύο θέματα που ε, σημειώνει στο σχέδιο εκθέσεώ του ο εισηγητή για την πρόοδο τη Μακεδονία, δηλαδή το 2010. Το σχέδιο εκθέσεω περιλαμβάνει σημαντικέ συστάσει, τι οποίε θα λάβουμε σοβαρότατα υπόψη μα ω κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιποι θεσμοί μα και βεβαίω και η απήχηση στον τύπο δείχνει το ενδιαφέρον που έχει το κοινό μας για, τις, για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας. Αφενός η κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Μακεδονία θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία νέων μίντια αλλά υπάρχει και μείγμα ε, δημοσίων και ιδιωτικών. Η κυβέρνηση μεταφέρει στην νομοθεσία τι ισχύουσε αρχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κυριότητα στα μέσα ενημέρωση και για την πρόσβασή του στην αγορά. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εργάζονται ελεύθεροι από οποιασδήποτε πιέσει και παρεμβάσει. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε χρήση των media outlets για συγκαλυμμένε επιχειρησιακέ, επιχειρηματικέ μάλλον ε, ατζέντε και ζητούμε να αποφεύγουν οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. η διαφανής κυριότητα των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης μια σημαντική ε, ανησυχία τη κυβέρνηση. Θέλουμε επίσης να συζητήσουμε μαζί σας και την πρόοδο που έχει γίνει στα θέματα της δικαιοσύνης για να εξασφαλιστεί ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί την προσπάθεια του εξυγχρονισμού του νομικού πλαισίου και της εφαρμογής του. Σχετικά με την δημόσια διοίκηση, η κυβέρνηση ήδη έχει υιοθετήσει τη νέα στρατηγική για την κατάστρωση των νέων αναγκών της διοίκησης, των απαιτούμενων προσόντων για την πρόσληψη των διαφόρων προσώπων και επίσης τα όσα έχει ζητήσει η αρμόδια υποεπιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κάνουμε και πρόοδο προς την λειτουργία πλήρους οικονομίας της αγοράς με οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα προσφέρουν μακροοικονομική σταθερότητα, χαμηλό πληθωρισμό και ε, ξεκάθαρες δημοσιονομικές πολιτικές ακόμα και μέσα σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Θα επιτύχουμε κατά πάσα πιθανότητα σημαντική η οικονομική ανάπτυξη το 2011. Μένουν βέβαια πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Η μακεδονική κυβέρνηση, ο τρόπος που αντιμετώπισε την κρίση δείχνει ότι έχει την δυνατότητα να προχωρήσει. Σήμερα ήλθαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταλλάξουμε απόψεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Μακεδονίας. Πολλοί εξημών που είστε παρόντες εδώ σήμερα γνωρίζετε πόσο εκτιμούμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήλθαμε επίσης να ζητήσουμε και την υποστήριξή σας για το επόμενο στάδιο της πορείας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έναρξη δηλαδή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το κοινό, το μακεδονικό κοινό θεωρεί το Ευρωπαϊκό, Σύμβολο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ως μέγα σύμβολο ανεξαρτησίας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Και ελπίζουμε ότι θα στηρίξετε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμφανιστεί ως ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ενταξιακής πορεία της Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Χατζημαρκάκη να μιλήσει για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα εκφράζω την ικανοποίησή μου που βλέπω πάλι τον ε, αναπληρωτή Πρωθυπουργό ο οποίος συχνά ε, προσέρχεται στις Βρυξέλλες, ο οποίος στα Σκόπια πάντοτε μας έχει ανοίξει όλες τις πόρτες. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα λοιπόν. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά η μεικτή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους φίλους μας στη Σομπράνγε και μαζί με τον Ζόραν Τάλερο, ο οποίος θα λάβει το λόγο μετά από μένα. Πάντοτε βρήκαμε ανοιχτέ τις πόρτες και μπορέσαμε να μιλήσουμε ανοιχτά για όλα τα προβλήματα που σημειώνονται. Πρώτα όμω θα ήθελα να σα συγχαρώ κύριε Αναπληρωτή, ε, κύριε Αναπληρωτά Πρωθυπουργέ. Όπως είπατε η οικονομική πορεία τη χώρα σα είναι υποδειγματική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Παρόλη την οικονομική κρίση η οποία έπληξε πολύ βαριά κυρίω τον νότιο γείτονά σα, μπορέσατε παρόλε τι διασυνδέσεις και διακλαδώσει των οικονομιών σα, μπορέσατε να αποσυνδεθείτε κατά κάποιο τρόπο και να συνεχίσετε την πορεία σας προς τα εμπρός. Πραγματικά υποδειγματικό υποδηματικός ο ρόλος σας για ολόκληρη ε, την περιοχή. Βέβαια, το ζήτημα, το διμερές ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί οδηγεί και συγκρούσεις και μέσα στην χώρα σας και προφανώς και ανάμεσα στις εθνι, εθνοτικές ομάδες και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αλβανική μειονότητα, αν μπορεί κανείς να την αποκαλέσει μειονότητα. Αυτό είναι κάπως ανησυχητικό, διότι όπως είπατε και εσείς φέτο είναι η δεκαετή επέτειο τη Συμφωνία Πλαισίου τη Οχρίδας και θα θέλαμε πολύ η κυβέρνησή σας, μάλιστα αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει μαζί σας, ότι ο πρόεδρός σας θα προσκαλέσει μεταξύ άλλων και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως και θα βρείτε βεβαίω παρά το πλευρό σα όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι και το Συμβούλιο αλλά και ιδίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σα υποστηρίξουν και θα είναι παρόντα τα όργανα αυτά, γιατί αυτή η δεκαετή επέτειο τη Συμφωνία Οχρίδα είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντική. Παρά τα, παρά συγχαρητήρια, θα έλθω και σε τρία θέματα τα οποία επέπεσαν στην αντίληψή μας και στις τελευταίες μας συνομιλίες. Πρώτο, η μεταχείριση του πρέσβεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερμάν Φουερέ, ο οποίος δεν είναι πλέον πρέσβης, συνταξιοδοτήθηκε προ λίγων εβδομάδων, αλλά δεν τον αποχαιρέτησε κανείς επισήμως, ενώ υπήρξε από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για την εξασφάλιση της ε, πορείας της χώρας σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προσευλήθη βαριά από βουλευτές του κόμματός σας, δεν, όπως είπα, τον απεχαιρέτησε επισήμως κανένας. Απευθύνω ωστόσο θερμό χαιρετισμό στον κύριο Φερέ σήμερα που είναι παρόν εδώ. Το θέμα της ελευθερίας του τύπου το θίξατε εσείς ο ίδιο. Ο Ζόραν Τάλερ νομίζω θα επανέλθει σε αυτό. Το τρίτο ωστόσο θέμα είναι ο πολιτικός διάλογος. Προφανώς επίκυνται νέε εκλογέ στην χώρα σας. Εμείς, εμάς μας ικανοποιεί το ότι πρόκειται να γίνουν πρόορες εκλογές. Δεν είμαστε όμως βέβαιοι εάν αυτό θα οδηγήσει σε, ε, σε κάποιο καθυσυχασμό της κατάστασης. Θα θέλαμε να μας προσκαλέσετε και ως μεικτή αντιπροσωπεία και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας προσκαλέσετε να συμμετάσχουμε στο γίγνεσθε της, ε, των εκλογών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάλερ, εισηγητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ε, ευκαιρία που μας δίνετε κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ για συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά το ότι βρίσκεστε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι έχουμε τακτικές επαφές. Ε, η Μακεδονία δεν είναι αρκετά παρούσα στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας για την επικοδομητική συνεργασία σας ε, με τις δραστηριότητές μας και να τονίσω ότι τον ίδιο στόχο έχουμε ο στόχος είναι κοινό. Η Μακεδονία το συντομότερο δυνατό να καταστεί μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση, αυτή είναι η θέση και τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και αυτό φαίνεται από το πρώτο σχέδιο του ψηφίσματο για τη Μακεδονία. Το Κοινοβούλιο ε, από όλες τις πολιτικέ ομάδε υποστηρίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων ενταξιακών με τη Μακεδονία και αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό. Γενικά όμως τις συζητήσεις για το ψήφισμα ανέκυψε ότι επικρατεί μεγάλη συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων και αυτό θα ανακύψει και από τις ε, ε, συζητήσεις μας σήμερα αναφορικά με τις 14 συμβαστικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το πρώτο ε, σχέδιο ψηφίσματος. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω το εξής, ότι όσοι παρακολουθούμε τις σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μακεδονίας, μεταξύ ΙΠΑ, Ουάσιγκτον και Μακεδονίας, Όσοι παρακολουθούμε λοιπόν αυτές τις ε, σχέσεις ε, διαπιστώνουν μια ευρεία συνένεση. Αφενός διαπιστώνουμε ότι πολλά έχει πετύχει η Μακεδονία όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά ε, την τελευταία 20 ετία της ανεξαρτησίας της. Αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Κατά πόσον για παράδειγμα η πρόοδος αυτή, η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά θετική και αρκετά γρήγορη. Να αναφερθώ στον πολιτικό διάλογο, το αναφέρετε και εσείς άλλωστε. Κατά δεύτερον, οι διεθνικές ε, σχέσεις, οι διεθνωτικές σχέσεις στο εσωτερικό της Μακεδονίας, το θέμα του δικαστικού συστήματος και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο όσο πιο δυνατόν ακριβές για την ευρωπαϊκή Εντάξει, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέλαμε ένα σαφές σχέδιο από πλευρά της κυβέρνησής σας και από το Κοινοβούλιο σας για το πώς σκοπεύετε να πετύχετε το στόχο της ένταξης. Κάποιες διευκρινήσεις επίσης να ζητήσω για την τρέχουσα κατάσταση ως προς τον πολιτικό διάλογο στη χώρα σας και να ρωτήσω τι προβλέπετε για τους επόμενους μήνες και σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και των δικαστηρίων. Επίσης, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε ως προς την 15 η επέτειο Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας και πώς σκοπεύετε να εξαλείψετε τα εμπόδια που μας αποτρέπουν από το να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ένταξης. Να ρωτήσω Επίσης, σε ποια φάση βρίσκεται η δίωξη κατά της Ελλάδα στο Διεθνές Πενικό Δικαστήριο στην Χάγη. Πού βρίσκεται αυτή η δίωξη, η κατάσταση. Θα πρέπει να περιορίζουμε το χρόνο ομιλία σε 1,5 λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γιαννάκου ζήτησε να μιλήσει. Σας δίνω το λόγο, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον αναπληρωτή ε, Υπουργό για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, για τις τοποθετήσεις του και ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις που δίνουν κάποιες ελπίδες να διευθετηθεί το θέμα που έχει ανακύψει με ένα κράτος μέλος. Ε, γιατί βεβαίως αυτό δεν είναι περίεργο, είναι αρκετά συνηθισμένο σε περιπτώσεις έναρξης διαπραγματεύσεων ένα κράτος μέλος να έχει αντιρρήσεις. Είχαμε το παράδειγμα άλλωστε της Σλοβενίας με την Κροατία ε, όμως πού βασίζεται αυτή η ελπίδα ε, κύριε Υπουργέ όταν ε, υπάρχει πρόταση από τα Ηνωμένα Έθνη όπως ανέφερε ο ίδιος ο Μπαν Μουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που το επισκέφθηκε την οποία η Ελλάδα δέχτηκε και εσείς όχι. Δηλαδή επειδή καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να πιεστεί ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις πριν διευθετηθεί το όνομα του ονόματος. Τι σκοπεύετε να κάνετε, διότι το πρόβλημα είναι σε εσά. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει σε γεωγραφικό προσδιορισμό και σύνθετη ονομασία. Επομένως τα πράγματα είναι συγκεκριμένα πια, δεν είναι στο θεωρητικό επίπεδο. Είναι πρακτικά και άμεσα. Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησής σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Ε, έχω μια αίσθηση ότι μας παρουσίασε μια εξειδανικευμένη εικόνα της κατάστασης στη χώρα του γιατί παρακολουθώντας και τον τύπο και τα γεγονότα εκεί βλέπουμε ότι τα πράγματα σε πολλά επίπεδα δεν πάνε στη θετική κατεύθυνση. Η ανεξαρτησία του τύπου πλήττεται κατάφορα, κάθε κριτική φωνή στην κυβέρνηση φημώνεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τίθενται ένα αμφιβόλο και ο πολιτικός διάλογος έχει παγώσει. Και από ό,τι παρακολουθούμε όλη η συζήτηση στη χώρα περιστρέφεται γύρω από πρόορες εκλογές και ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει κηρύξει στάση εργασιών. Αν σε όλα αυτά προσθεθούν ε, και γεγονότα και προσωπικές επιθέσεις από αξιωματούχους εναντίον του Αμερικάνου πρέσβη, του κύριου Φουερέ ή από ορισμένου κύκλους και εναντίον του ίδιου του εισηγητή του Κοινοβουλίου του κύριου Τάλερ, το κλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι αρνητικό. Ο κύριος Γκρουευσκής συχνά προσπαθεί να πείσει ότι φταίει η Ελλάδα για αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Ε, νομίζω ότι η Ελλάδα εχει διαμορφωθει στη χωρα νομιζω αναλάβει τις ευθύνες της, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει επανειλημμένως πρωτοβουλίες και με τις διμερείς επαφές στην κατεύθυνση εξέβρισης λύσης ε, καλό θα ήταν και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο κύριος γκρούευσκι να αναλάβει πρωτοβουλίες σε μια προοπτική επίλυση, ώστε να αποδείξει ότι πραγματικά τον ενδιαφέρει η επίλυση της διαφοράς και άρα η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλημέρα σας, κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών μας ομάδων θέλει να προσχωρήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι πολίτες της Μακεδονίας να καταστούν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε αυτή η πορεία σας να οδηγήσει προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μου σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση, εθνοτική συνεννόηση πριν από τις εκλογές και να ορίσετε και το θέμα της αυτοδιάθεσης. Δυστυχώς βλέπουμε τώρα τελευταία ότι οι κάτοικοι της Μακεδονίας που θεωρούν ότι προέρχονται από τη βουλγαρική μειονότητα την χάνουν απαράδεκτης μεταχείρισης από τους δημόσιους φορείς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μην επιδεινωθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε, να μας δώσετε τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στις ε, μυστικές υπηρεσίες της χώρας σας, πού βρισκόσαστε ως προς τη σχέση σας με τη Σερβία και τα αρχεία που βρίσκονται στο Βελιγράδι. Επίσης, θα ήθελα να ε, βελτιωθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας και με τις άλλες χώρες, δηλαδή τη Βουλγαρία και την Ελλάδα δεχόμενη την ιστορία τους και μη προβαίνοντας σε δόλιους χειρισμούς. Ελπίζουμε να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, καταρχά θα ήθελα να σα καλωσορίσω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τα θετικά στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσατε. Να πω όμως και κάποια λόγια τα οποία ενδεχομένω ε, να μην σας ευχαριστήσουν. Πριν από κάποιες ημέρες έλαβαν κάποιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου μία επιστολή από έναν απελπισμένο νεαρό, ο οποίος ε, έγραφε με τις δικές του λέξεις, με το δικό του στυλ αν θέλετε, πώς ε, έχει η κατάσταση στη χώρα σας. Και νομίζω ότι η επιστολή αυτή μας προκαλεί αρκετές ανησυχίες. Ε, καλό θα ήταν να δώσουμε προσοχή, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνει την ε, γνώμη της πλειονότητας των νέων. Να μην φοβόμαστε τη λέξη της κόπωσης της ε, διεύρυνσης. Όχι, κοιτάξτε, η διεύρυνση αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς το σεβόμαστε αυτό στο έπακρο. Νομίζω ότι για την επίλυση ανοιχτών ζητημάτων θα πρέπει να επιδείξετε με πιο μεγάλη ευελιξία, λιγότερο εθνικισμό, λιγότερη αν θέλετε προσκόλληση στην ιστορία και πιο ε, μεγάλη ανησυχία για τα συμφέροντά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμστορφ λέει ο πρόεδρο είναι ο τελευταίο που θα μιλήσει, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Όχι, όχι, θα μιλήσετε. Είσαστε στον κατάλογο ομιλητών, αλλά θα θέλαμε στο σημείο αυτό να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Και τώρα θα είμαι και πιο αυστηρός, γιατί θα γίνει η συζήτηση για την Μακεδονία και πιο μετά. Ο κύριος Κούκαν, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο οικοδομητικό διάλογος με την Μακεδονία. Τρεις ερωτήσει έχω να σας απευθύνω. Πρώτα, η πολιτική κατάσταση πριν από τις εκλογές. Όπω ξέρουμε, τα σοσιαλιστικά κόμματα μποϊκοτάρουν το κοινοβούλιο. Αυτό φυσικά είναι απαράδεκτο. Και επιπλέον απειλούν ότι δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Χτες ανακοινώθηκε ότι ο Πρωθυπουργός θα συναντιόταν με τον ε, αρχηγό της αντιπολίτευσης για να συζητήσει τέτοια θέματα. Τι θα γίνει λοιπόν, θα συμμετάσχει, δεν θα συμμετάσχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις εκλογές και τι θα γίνει και με την προετοιμασία του εκλογικού κώδικα. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Και μια τρίτη ερώτηση για την συμφωνία της Οχρίδας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό έχει αποδειχθεί και από τον ε, χρόνο που έχει περάσει. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής. Πώς λοιπόν θα γιορτάσετε την επέτειο αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριε Πόσελτ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος εκεί πίσω μίλησε για εθνικισμό. Ο εθνικισμός δεν αποτελεί προνόμιο των υποψήφιων χωρών. Εθνικισμό υπάρχει, εθνικισμός υπάρχει και στα, στις χώρες μέλη. Και ο εθνικισμός είναι αυτός που μπλοκάρει να γίνουν αυτά τα οποία η συνάδελφος Γιαννάκου δικαίως ανέφερε και έχει χάρηκα που εξ αρχής μίλησε για διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε με σαφήνεια ότι θέλει να ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Ουγγρική Προεδρία την προηγούμενη εβδομάδα απάντησε σε μια ερώτηση και δήλωσε ότι ελπίζει υπό τη διάρκεια της Προεδρίας της να ξεκινήσει η σύσταση της Επιτροπής για έναρξη των διαπραγματεύσεων. Να ρωτήσω λοιπόν τον απληρωτή Πρωθυπουργό αν ε, το επιθυμούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν ξεκινάει η διαδικασία αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα μπλοκάρισμα, αλλά υπάρχει και μια ενδιάμεση συμφωνία. Πείτε μου λοιπόν, γιατί αυτή η ενδιάμεση συμφωνία στη συζήτηση δεν διαδραματιζεί κανένα ρόλο. Και μια πολύ μικρή προσωπική παρατηρήση, κύριε Χατζημαρκάκη, δεν νομίζω ότι είναι εντάξει το γεγονός ε, ότι ξεκινάμε εδώ μια συζήτηση για τον κύριο Φουερέ, γιατί έχω διαφορετική άποψη για τον κύριο Φουερέ, αλλά για λόγους δικαιοσύνης δεν μπορώ να την εκφράσω, γιατί δεν θεωρώ ότι εδώ είναι ο τόπος να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Θέλω να μοιραστώ μερικές σκέψεις και ορισμένες ερωτήσεις μαζί σας. Η χώρα σας, έχει με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Βρίσκεται λοιπόν κυριολεκτικά στο κατόφλι της ευρωπαϊκής πόρτας. Και πρέπει να σας πω ότι ιστορικά, και το γνωρίζετε άλλωστε, στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας είχαν χώρες με σταθερές, όριμε και λειτουργούσε δημοκρατίε. Εδώ και πολλού μήνε όμω η χώρα, σα χώρα σας ταλαιπωρείται με αδυναμία μια αποτελεσματική προετοιμασία, μια πρόορη όπω όλα δείχνουν εκλογική αναμέτρηση. Η αντιπολίτευση δεν συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Χωρί αντιπολίτευση επιχειρείται να εκλεγεί πρόεδρο τη εκλογική επιτροπή, Εκλογικοί κατάλογοι αμφισβητούνται. Ο καθορισμός των εκλογικών περιφερειών βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο και σε απόλυτη εκκρεμότητα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται επίσης ο καθορισμός της διαδικασίας για την ψήφο της Διασποράς και η χθεσινή πολύ και δραματική συνάντηση Γκουρεύσκη και Τσεβερκόφσκη δεν παρήγαγε οποιοδήποτε αποτέλεσμα για να λύσει το πρόβλημα αυτό. Και ουδής γνωρίζει τι θα γίνει και κανείς δεν, προβλέπει, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Για όλα αυτά που αναφυσβήτητα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή σας πορεία φταίει η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και να του πω ότι μπορεί να θεωρηθείτε ε, λαϊκιστής για πολλούς λόγους γιατί υπάρχουν αυτές οι πρακτικές ακόμα και σε ορισμένα κράτη-μέλη και σε κράτη-μέλη. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξής. Για τον ευρωπαϊκό σας ε, δρόμο θα πρέπει να δείτε πώς θα ορίσετε το, τον ανθρωπιστικό παράγοντα και θα πρέπει να δεχτείτε το γεγονός ότι θα πρέπει να έχετε μεγάλες μεγάλη απόδοση στον δημόσιο τομέα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι δράσεις σας έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η πολιτικοποίηση του δημοσίου τομέα. Ο κύριος Τάνοκ, παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και από την ομάδα του ECR και ως κοιόδης για την έκθεση της Τάλλαρης. Διαφωνώ με τον κύριο Τάλλαρη γιατί ήταν εξαιρετική η έκθεση του, αλλά αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την... Μάλλον δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεπαρκή παρουσία της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, κάνει πολύ έντονες προσπάθειες η, η κυβέρνησή σας και διαπιστώνουμε ότι και εσείς και ο Πρωθυπουργό σας συμμετέχετε σε διάφορες εκδηλώσεις ε, στο Κοινοβούλιο και αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για την προώθηση των συμφερόντων σας. Ε, επίσης, να συγχαρώ την κυβέρνησή σας για τις προσπάθειές της ε, σε μια δύσκολη στιγμή και λυπάμαι για το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου από την, το κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα σας και εγώ όπως και άλλοι ομιλητές λυπούμε ε, για το ότι δεν μπορεί να επιληθεί το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα και προφανώς ε, και χαίρομαι που τώρα για παράδειγμα ε, προσελκύεται άμεσες ξένες επενδύσεις και από την χώρα μου και θεωρώ ότι με την έλλειψη γραφειοκρατίας και με το καλό επενδυτικό περιβάλλον ε, είναι καλέ οι προπτικές για τη χώρα σας. Και εγώ ανησυχώ για την σταθερότητα της συμφωνίας τη ΟΧΡΙΔΑ και με ανησύχησε στη χώρα σας η... το δυναμικό ε, μεταξύ Αλβανών για παράδειγμα και νομίζω ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξη και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα. Ο κ. Κυρίλοφ παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκεται μαζί μας εδώ ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό κ. Ναουμόφσκι και να πω ότι υποστηρίζω μία σειρά συναδέλφων που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ε, το συντομότερο δυνατόν να αναφέρω το θέμα του πολιτικού διαλόγου με ένα παράδειγμα. Κύριε Νομόφσκι, ε, υπάρχει αυτό το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και χαρήκαμε όταν αποφασίστηκε να ε, συμμετέχει και να ηγηθεί η αντιπολίτευση του Συμβουλίου. Φαίνεται όμως ότι δεν λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες, λαμβάνουν πολύ περιορισμένε πληροφορίες για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης της χώρας σας. Ισχύει αυτό και γιατί. Και ανησυχώ, όπως και ο εισήγητης ο κ. Στάλερ θεωρώ ότι αρνητικό είναι το εξής. Από τη στιγμή που κάποιος ε, επιδεικνύει κριτικό πνεύμα για κάποια θέματα, κατευθείαν αντιμετωπίζει αντιδράσεις. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να συζητηθεί αυτό τώρα, αλλά ξέρετε, ο προσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Όπως είπαν και πολλοί άλλοι, να υπενθυμίσω δύο θέματα θα ήθελα. Η Μακεδονία είναι η χώρα η οποία βρίσκεται τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο ως χώρα υποψήφια. Και νομίζω ότι η κατάσταση αυτή ε, συνδέεται με έναν ε, πατριωτισμό ο οποίος ε, λανθασμένα γίνεται αντιληπτός στην Ελλάδα και νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει πέρα από τα κομματικά όρια ότι είναι προς το συμφέρον της όταν η Μακεδονία δεν θα προκαλεί διεθνικά προβλήματα τα οποία τα πασαλείψαμε με την Συμφωνία Πλαίσιο της Αχρίδας. Νομίζω λοιπόν ότι και η γειτονική χώρα θα πρέπει να έχει συμφέρον να μην να κλιμακωθούν τα προβλήματα αυτά και επιτέλους να λυθεί το θέμα του ονόματος. Και κατά δεύτερον οι σοσιαλιστές εμποικοτάρουν το κοινοβούλιο, το ξέρουμε αυτό και από την Αλβανία. Θα ήθελα να ξέρω ποια αφορμή χρησιμοποιούν οι σοσιαλιστές για να μποϊκοτάρουν το κοινοβούλιο. Έχει να κάνει με, την, ε, ε, με το κανάλι της τηλεόρασης το οποίο μεταχειρίζεται άσχημα η κυβέρνηση, υποτίθεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα, ο σταθμός αυτός δεν έχει πληρώσει φόρους. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμστορφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω γιατί εκτός της περιοχής αυτής ε, δεν υπάρχει κατανόηση για το θέμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο θέμα ε, του ονόματος και στον άτομο τα πράγματα θεωρούνται παρανοϊκά. Στο Λουξεμβούργο υπάρχει ε, μια χώρα, κοιτάξτε και στην, ε, στο Βέλγιο, μάλλον υπάρχει χώρα Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο υπάρχει και επικράτεια, ε, περιφέρεια που ονομάζεται Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχει αυτό πρόβλημα. Αυτό που αναφέρεται στο συμβαστικό, στη συμβαστική τροπολογία 5 είναι η κουλτούρα συμβιβασμού που επικρατεί στη χώρα. Η Αλβανία δεν έχει λάβει καθεστώς ενταξιάκή χώρας λόγω της επιδείνωσης του πολιτικού διάλογου. Και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την πολιτική αυτή κουλτούρα. Ισχύει, κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, ότι ο κύριο Ταλέσκη, δήμαρχος του Πίτελα, είχε συνδέσει και είχε κάνει συγκρίσεις μεταξύ ε, των, ε, της πολιτικής των ε, Ναζί με την πολιτική των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω ε, ομαδοποιημένα γιατί αφορούσαν ε, τα ίδια θέματα. Κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Φουρέ, τον πρώην πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσω από τον κύριο Χατζημαρκάκη να σας υπενθυμίσω ότι αντίθετα από το ότι θεωρείται ότι δεν υπήρξε σωστός αποχωρισμός, ε, υπήρξε ε, δεξίωση από το Κοινοβούλιο, από τον Πρωθυπουργό, από εμένα. Σε όλες ε, τις συναντήσεις με τον πρεσβευτή εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη μας για την συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα και είμαστε βέβαιοι ότι και στις μελλοντικές δραστηριότητές τους θα παραμείνει δεσμευμένος για την ατζέντα αυτή. Ήταν στη χώρα μας για πέντε χρόνια και παραπάνω και κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτή θεωρήσαμε ότι πέρα από κάποιες κριτικές ήταν θετικός ο τρόπος ε, που αναφέρθηκε και εν πάση περιπτώσει και οι κριτικές αυτές είχαν θετικό σκοπό για τον πολιτικό διάλογο. Αληθεύει ότι η θέση, ότι η αντιπολίτευση, συγγνώμη, μποϊκοτάρει το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και ακριβώς αυτή η κατάσταση είναι που προκαλεί τις εκλογές για το 2011 δεν υπάρχει υποψήφια χώρα ή χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει το Κοινοβούλιο και επειδή μέλο τη χώρας μας συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε πρόορες εκλογές. Μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην πολιτική μας πρακτική και η κυβέρνηση έχει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο συμφώνησε να διεξαχθούν πρόορες εκλογές. Έγιναν χτες συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο ε, κομμάτων, διήρκησαν 10 ώρες και τέθηκαν από την αντιπολίτευση, ε, μάλλον έγιναν αποδεκτές 30 30 αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στο Κοινοβούλιο σήμερα θα, ελεχθεί, θα εκλεχθεί ο πρόεδρος της εκλογικής ε, Επιτροπής και ελπίζουμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα συμπεριλαμβανημένες της αντιπολίτευσης παρά το γεγονός ότι έχουν μόνο 18 από τους 120 βουλευτές θα αναλάβουν τις ευθύνε τους. Να ευχαριστήσουμε όλους τους βουλευτές που εξέφρασαν την ανησυχία τους και που ζήτησαν από την αντιπολίτευση να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλδημοκρατών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όσο προχωράμε προς την ολοκλήρωση των ε, θεμάτων της ατζέντα που έχουμε συμφωνήσει, θα μπορέσουμε να περάσουμε σε προώρες εκλογές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και μετά ελπίζουμε ότι τα μέλη της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν να μποϊκοτάρουν το Κοινοβούλιο επειδή όπως ξέρετε όλοι οι βουλευτές έχουν εκλεχθεί προκειμένου να εκπροσωπούν το εκλογικό τους, την εκλογική τους περιφέρεια στο Κοινοβούλιο κάποιες ερωτήσεις για τη Συμφωνία Πλαίσια της Οχρίδας. Να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και αποτέλεσε ένα υπόδειγμα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων ε, στα Βαλκάνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Μακεδονία έχει τα ίδια πρότυπα για, για τις μειονότητες όπως η Σουηδία, αλλά να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Μακεδονία είναι η Σουηδία των Βαλκανίων σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την σωστή εκπροσώπησή τους στη δημόσια διοίκηση, τη χρήση των γλωσσών, σωστή αντιπροσώπευση στο δικαστικό σώμα, στο αστυνομικό σώμα, σε άλλους θεσμούς, σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεων, στο κοινοβούλιο, στις τοπικές κυβερνήσεις. Άρα θεωρώ ότι αποκινούμε όλους τους εκπροσώπους από όλα τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και αυτούς που εκπροσωπούν τις κοινότητες και τις ε, μειονότητες, θα περάσουμε στην αρτασμό της ε, επαιτίου της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας και ο πρόεδρος της χώρας ε, έχει προγραμματίσει να συμμετάσχει σε κάποιες εκδηλώσεις σχετικές. Τονίζουμε τη σημασία της συμφωνίας αυτής και εξακολουθούμε να αν διακηρύττουμε το πνεύμα της συμφωνίας και σε τοπικό αλλά και σε κρατικό επίπεδο. επρόκειτο για μια συμφωνία με πλεονεκτήματα για όλες τις κοινότητες, όχι μόνο για τις μειονότητες. Και χαιρόμαστε που ως τώρα δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να κινούμαστε και στο μέλλον. Κάποιες ερωτήσεις τώρα τέθηκαν για το θέμα του ονόματος και τα σχέδια ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μας έθεσε η κυρία Γιαννάκο, ο κύριος Κουμουτσάκος, η κυρία Κοπά. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η πρόθεση της κυβέρνησης Μακεδονίας είναι να συνεχίσει να αναζητά μία αμοιβαία αποδεκτή λύση ακριβώς επειδή πρόκειται για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ευρωτελική μας ενοποίηση η οποία διακυβεύεται κατά την αναβολή της επίλυσης του θέματος και εμείς ε, ε, θέλουμε να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση, μια λύση συμβιβαστική. Όταν λέμε συμβιβαστική, ε, εννοούμε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις και των δύο λύση, η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τη θέση της μίας πλευράς, δεν αποτελεί συμβιβαστική λύση. Άρα μια συμβιβαστική λύση η οποία λαμβάνει 100% της υπόψη της θέσης μιας πλευράς δεν μπορεί να θεωρηθεί τη συμβαστική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το λαό της Μακεδονίας. Είναι πρόθεση της κυβέρνησής μας να αναζητήσει μια λύση μέσω ειλικρινούς διαλόγου μαζί με την Ελλάδα και θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι η χώρα η οποία θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ενοποίηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ακριβώς επειδή πρόκειται για το πιο παλαιό κράτος μέλος της περιοχής και επειδή σημαντικά έχει ωφεληθεί από την αρχή της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επιδείξει τέτοιο πνεύμα και προς τις άλλες χώρες της περιοχής. Θεωρούμε επίσης ότι η ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι προς συμφέρον και της Ελλάδας και από κοινού με την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να επικεντρωθούμε στις πολιτικές της ε, περιοχής μας σε 30-50 χρόνια οι χώρε μα θα εξακολουθήσουν να είναι φυσικά γειτονικέ χώρες και θα πρέπει από κοινού να εργάζονται για το κοινό συμφέρον ε, των πολιτών μας. Αναφέρθηκε η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 από τον κύριο Πόσελτ όταν συμφώνησε η Δημοκρατία της Μακεδονίας να αλλάξει την εθνική της σημαία. Αφετέρου η Ελλάδα συμφώνησε να μην μπλοκάρει την ένταξη ε, της χώρας μας σε διεθνείς οργανώσεις. Η συμφωνία αυτή ε, υπεγράφει από τον κύριο Παπούλια, ο οποίος είναι πρόεδρος σήμερα της Ελλάδας, ήταν τότε υπουργό και θεωρούμε ότι η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι είχε υπογραφεί τότε. Ε, ήμασταν μάρτυρες των ενεργειών της γειτονική μας χώρας το 2008 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που δεν ήταν απόλυτος συμμορφωμένες με τις με τη συμφωνία Πλαισίου της Αχρίδας και γι' αυτό λοιπόν υποβάλαμε δίωξη στο δικαστήριο. Αναμένουμε ότι θα αρχίσει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα η δημόσια ακρόαση. Σύμφωνα με τις πρακτικές του δικαστηρίου, η απόφαση θα ε, βγει κάποια στιγμή μέσα στο έτος. Όποια και αν είναι η απόφαση που θα λάβει το δικαστήριο, δεσμευόμαστε να την εφαρμόσουμε και το ίδιο περιμένουμε και από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για μία υπόθεση η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να σχολιάσουμε περαιτέρω μέχρι ότου ολοκληρωθεί η δικαστική εξέτασή της. Κάποιες ερωτήσεις τώρα για την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης. Επιτρέψτε μου να σας ε, υπενθυμίσω, όπως έχω πει και στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια ε, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν πλέον ε, νέα μέσα στη χώρα, ηλεκτρονικά μέσα, έντυπα μέσα, και όπως αναφέρεται στο σχέδιο ψηφίσματος, μας ε, ανησυχούν και εμάς ε, ε, θέματα αδιαφάνειας ως προς την ιδιοκτησία μέσων. Έγιναν κάποια, μάλλον κάποια περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων προκάλεσαν ανησυχία στο ευρύ κοινό. Να σας υπενθυμίσω ότι στη Μακεδονία, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες, όλες οι πολιτικές οντότητες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν φόρους στη χώρα όπως και όλοι οι πολίτες. Η εφορία τα τελευταία πέντε χρόνια έχει κάνει ελέγχους σε περισσότερες από 90 οντότητες ε, που ασχολούνται με διαδικασίες και ε, με τα μέσα ενημέρωσης είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή και ανακάλυψε ε, ατασταλίες φορολογικές οι οποίες προκάλεσαν πρόστιμα. Δύο εθνικά κανάλια τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 300.000 ε, ευρώ το ένα κανάλι, 200.000 ευρώ το άλλο κανάλι. Δεν υπήρξαν οποιασδήποτε ενστάσεις εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ατασταλίες ε, φορολογικές και συνεχίζονται, συνεχίζονται και άλλοι έλεγχοι. Να σας υπενθυμίσω ότι η μακεδανική νομοθεσία έχει τους ίδιους, ε, ε, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και το γερμανικό δίκαιο για τη φορολογία και επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση Τάξου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τακτικά ενημερώνεται για τις δραστηριότητε μας, για τις δραστηριότητες της μακεδονικής εφορίας και των ελέγχων που λαμβάνουν χώρα στα μέσα ενημέρωσης. Έγινε και έλεγχο σε μία από τις εθνικές τηλεοράσεις ε, τις τελευταίες εβδομάδες και τα τελευταία δεδομένα υποδεικνύουν ένα ποσό 9 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια ως προς φορολογικές ατασφαλίες. Θεωρούμε ότι αν και πρόκειται ε, για μέσο ενημέρωσης, παρόλα αυτά πρέπει να πληρώνει τους φόρους του. Και ότι εκόπη η εκπομπή των προγραμμάτων καμία ημέρα. Ως κυβέρνηση δεσμευόμαστε να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα και τη φοροδιαφυγή. Καταπολεμούμε επίσης και την διαφθορά. Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθεί κανείς από τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Αν πρόκειται δηλαδή για μια ε, νομική οντότητα με ε, λειτουργία μέσου ενημέρωσης. θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που θα εκδοθούν από το δικαστήριο αν το ζητήσει και η κυβέρνηση. Τέθηκε θέμα παγώματος λογαριασμών μιας νομικής οντότητας εθνικού καναλιού τηλεόρασης. Να σας υπενθυμίσω ότι το πάγωμα του λογαριασμού αποτελεί τμήμα του νόμιμου συστήματος και της νομοθεσίας των πιο πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο λοιπόν μπορεί να αποφασίσει να παγώσουν λογαριασμοί όπως ε, στη Μακεδονία όπως και σε πολλές άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πάγωμα των λογαριασμών αποτελεί ένα τμήμα, ένα μέρος των ε, δυνατοτήτων του δικαστηρίου. Επίσης αναφέρθηκαν Κάποιες ερωτήσεις έγιναν για τις σχέσεις καλής γειτονίας από τον κύριο Κοβάτσεφ και από άλλους συναδέλφους. Η Μακεδονία δημόσια έχει διακηρύξει πάσα πρόθεση να συνεχίσει την οικοδόμηση καλών σχέσεων με όλους τους γείτονες, με συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, του Κωσυφοπεδίου. Είναι η μοναδική χώρα στην περιφέρεια η Μακεδονία που δεν έχει ε, ζητήματα, δεν αντιμετωπίζει ζητήματα ε, συνοριακά, συνοριακών διαφωνιών. Και σε πολλές περιστάσεις δηλώσαμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών να συνεχίσουν την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε βάθος για πιο οικοδομητικές σχέσεις, ιδιαίτερα με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα. γιατί μας συνδέουν πολλά και με την Ελλάδα και με την Βουλγαρία και αυτά θα πρέπει να τονίσουμε για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Τέθησαν και κάποιες ερωτήσεις για την ε, διοίκηση. Η Μακεδονία όπως και όλες οι άλλες χώρες ε, που ήταν ε, τμήματα του πρώην κομμουνισμού. Τα τελευταία χρόνια έγιναν ε, εκτεταμένες προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση από το 2008 και 2009. Η κυβέρνηση ξεκίνησε και τραποποίησε ε, νόμους για την διοίκηση από κοινού με τους από την ΣΥΓΜΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εισαχθεί ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει οποιαδήποτε δυνατότητα πολιτικής επιρροής ε, στην διοίκηση. Αποτέλεσε αυτό προτεραιότητα της κυβέρνησης και έγινε και μια ειδική υπουργική συνάντηση μάλλον υπάρχει και ειδικό Υπουργείο που αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε να έχουμε όρατα αποτελέσματα. Έχουμε ένα πακέτο νόμων στην κοινοβουλευτική διαδικασία που θα επιτρέψει να γίνουν όλα τα μεταρρυθμιστικά βήματα λαμβάνοντας υπόψη και τις ανησυχίες των πολιτών. Επίσης, ε, θα προωθηθούν και οι προτάσεις ε, και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες ε, για την υποστήριξη όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμβάλει στην περιοχή αυτή. Then, uh, there were questions on the... Ανέκυψαν και ορισμένα ερωτήματα από τον κύριο Κυρίλοφ ως προς το Εθνικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα ήθελα να σας πω ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση για πρώτη φορά έγκαιρα αποστέλει πληροφορίες σε τριμηνιαία βάση στο Εθνικό Συμβούλιο και σε όλα τα άλλα όργανα με τις κατάλληλες πληροφορίες για την έγκριση της ε, νομοθεσίας Θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα δεν ε, είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί πολιτικά, αφορά όλες τις εθνικές ομάδες και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει από κοινού για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Δεν θα πρέπει να μολύνουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα με τη, την καθημερινή πολιτική ή μικροπολιτική. Ο κύριος Κουμουτσάκος υπέβαλε ένα ερώτημα, δηλαδή ε, κατά πόσο η Ελλάδα φέρει την ευθύνη για τα πάντα, κατά πόσο φταίμε εμείς, ποια είναι τα σχέδιά μας για ένα σύνθετο όνομα στο μέλλον, κατά πόσο φταίει ο δικός μας πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι στυλιτεύσαμε την Ελλάδα για όλα τα δεινά που, βρήκαν τη χώρα μας, αλλά ε, δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να αρχίσει η ενταξιακή πορεία και το ΝΑΤΟ κρίνει ότι πληρούμε όλες τις συνθήκες έτσι ώστε η χώρα μας να κληθεί να γίνει πλήρες μέλος και του ΝΑΤΟ. Ένα κράτος του ΝΑΤΟ αντιτάχθηκε στη συμμετοχή της χώρας μας και γνωρίζουμε ποια χώρα είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να την κατονομάσουμε εκ νέου. Προχωρήσαμε αρκετά σε αυτή την ε, ιστορία του ονόματος. Θα θυμόσαστε, αρχικά η Ελλάδα ζήτησε ένα σύνθετο όνομα ότι δεν πρέπει να καλούμεθα Μακεδονία, αλλά να έχουμε ένα σύνθετο ε, όνομα. Μετά σύνθετο όνομα με γεωγραφική μνήα και μετά στη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ προτάθηκε το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια αν και υπήρχε γεωγραφική μνήα όπως ζήτησε η Ελλάδα μετά, ζητήθηκε σύνθετη ονομασία με γεωγραφική μνήα η οποία να είναι άνω και μετά σύνθετη ονομασία με γεωγραφική μνήμα με τη μνήμα Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα από τα συμβαλόμενα μέρη ε, συμπτήσει τη λύση, δηλαδή την περιορίζει, περιορίζει τα περιθώρια λύσης. Η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτα δεν μιλάμε για ιστορία ή γεωγραφία ή για την ευρωατλαντική μας ε, ολοκλήρωση. Έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική κατάσταση. Κάποιος αναφέρθηκε στο Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Υπάρχει ευρύτερη περιφέρεια ε, Λουξεμβούργου και δεν υπάρχει καμία διένεξη μεταξύ Λουξεμβούρου και Βελγίου. Οι χώρες αυτές έχουν μια αγαστή συνεργασία και ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Αυτό, αυτό το πρότυπο θα πρέπει να ακολουθήσουν η Ελλάδα και η Μακεδονία για να άρουν οποιαδήποτε διμερή διαφορά στο βαλκανικό χώρο. Επίσης, μια άλλη υποψήφια χώρα είχε μία διμερή διένεξη με γείτονα χώρα, δηλαδή Σλοβενία και Κροατία. Ξέρουμε ότι η Σλοβενία έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία είναι μία υποένταξη χώρα και θα εξευρεθεί μία λύση για τη διμερή αυτή διένεξη. Εάν υπάρχει πραγματική θέληση και από τις δύο πλευρές, τότε θα το επιτύχουμε και εμείς. Η δημοκρατία της Μακεδονίας δεν είχε καμία πρόθεση να αναζητήσει κάτι το οποίο δεν μας ανήκει. Θέλουμε τα ίδια κριτήρια να ισχύουν όπως και για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προσπαθούμε να πληρούμε όλα τα κριτήρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις γείτονες χώρες να ανταποκριθούμε με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία έτσι ώστε να εντάξουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές στη... και για τη χώρα μας. Oh, uh, uh, Uh, Ως προς την ε, διαδικασία αυτή ελήφθη μία απόφαση να εγκρίνουμε αυτό το νόμο στον οποίο ε, προαναφερθήκατε εσείς. Θέλουμε να ε, διαλευκάνουμε, διαλευκάνουμε όλα τα θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα των κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών Ορισμένα αρχεία ε, ανήκαν στην, ε, στο Βελιγράδι, στην Ιν Σερβία, ήταν της ε, πρώην ε, Ιουκοσλαβικής Συνομοσπονδίας, Ομοσπονδίας, αλλά και οι δύο χώρες έκριναν ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα, δηλαδή θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και αρχεία. Could you say just briefly what you think of what Mayor Zaleski According to, to his words, κατά τα λόγια του την επόμενη μέρα ε, ο πολίτης αυτός ε, θεώρησε ότι λάθος αναφέρθηκαν τα λόγια του, δεν είχε καμία πρόθεση να καταφερθεί κατά του ολοκαυτώματος και του μνημείου που υπάρχει στα Σκόπια και ήταν λάθος από πλευράς ΜΜΕ αυτή η μνήμα. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση για το θέμα της ε, Μακεδονίας. Ναι, για 10 δευτερόλεπτα έχετε το λόγο. Αναφερθήκατε στην απόφαση του ΝΑΤΟ το 2008 όπου αναφέρθηκε ότι όλα τα κράτη-μέλη διαφωνούσαν με την θέση της Ελλάδας ή οι άλλοι διαφώνησαν με την Ελλάδα, άρα δεν ελήφθη απόφαση. Επειδή βρισκόμαστε λίγες ε, μέρες πριν από μια απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης, θα ήθελα να πω ότι η Συμμαχία έλαβε ομόφωνη απόφαση και δεν ήταν από το της ελληνικής θέσης ομόφωνα αποφάνθηκε ότι όταν επιληθεί το ζήτημα τότε η χώρα θα προσχωρήσει στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ήταν ομόφωνη απόφαση των χωρών του ΝΑΤΟ. Um, δεν υπάρχει όμως, δεν είναι μυστικό για το ποια ήταν η χώρα η οποία αντέδρασε. Αυτό που είπα είναι ότι όλες οι χώρες αναγνώρισαν ότι εκπληρεί τα κριτήρια για να εισχωρήσει για να ενταχθεί στην ε, Βορειοατλαντική Συμμαχία και υπήρχε βεβαίω ένα θέμα, το οποίο νομίζω γνωρίζουμε όλοι περί τίνος πρόκειται, το οποίο εμπόδισε την πορεία αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι για το ενδιαφέρον που δείξατε και για τις ερωτήσεις που υποβάλλατε. Θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα στη συζήτηση για τη Μακεδονία. It's a public debate, so you're welcome to stay. Okay. Okay. Yeah. Now, uh, colleagues, please, we have to continue. Να συνεχίσουμε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Θα συζητήσουμε τώρα πάλι την έκθεση για τη Μακεδονία, την έκθεση προόδου. Κύριε Τάλερ, εσείς. Mr. Έχει το λόγο, κύριε Τάλερ. Μην περιορίζετε να συνομιλείτε με τον κύριο Κούκαν, ενώ μπορείτε να τα πείτε σε όλους μας. Πόσο μου δίνετε, 10 λεπτά ή μία ώρα. Ας μπορέσουμε να τελειώσουμε τη συζήτηση ε, μέχρι τις 11.30. Τρία λεπτά λοιπόν για σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η ευκαιρία που είχαμε τώρα τη δυνατότητα να ακούσουμε και να συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο της κυβερνήσεως της Μακεδονίας και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με τη συζήτηση για το ψήφισμα περί Μακεδονίας. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες για το σχέδιο εκθέσεως. Πιστεύω απολύτως ότι μπορέσαμε με επιτυχία σε συνεργασία με τους κοιόδης συγητές να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή έκβαση, δηλαδή να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις, ε, στις συμβαστικές τροπολογίες όσο το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες των συναδέλφων μας. Και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσουμε το ίδιο το ψήφισμα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων για πλήρη ένταξη της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας Μακεδονίας αμέσως. Έχουμε δύο τέτοιε θέσει, δύο τέτοιε συστάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συζητούμε την πρόταση αυτή εδώ και καιρό. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα όπου προσπαθούμε να δώσουμε και κάποια μηνύματα στους ε, φίλους μας στη Μακεδονία. Και θα, του θα τους συμβουλεύσω και θα εκφράσω την ελπίδα να θεωρήσουν τις επιθυμίες αυτές ως μια ξεκάθαρη λίστα για το τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτούς, δηλαδή και σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης αλλά και για όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν όταν προσέρχεται και κρούει τις θύρες μας μια νέα χώρα. Δεν έχω επαρκή χρόνο τώρα για να συζητήσω με λεπτομέρειες τις συμβαστικές τροπολογίες. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν 14 συμβιβαστικές οι οποίες έχουν περιλάβει δεκάδες μεμονωμένων τροπολογιών και εγώ βεβαίως βάζω συν και σε πολλές άλλες τροπολογίες που έχουν πρόταθεί. Στην συμβιβαστική ένα επαναλαμβάνουμε ότι τα διμερεί θέματα πρέπει να επιληθούν με πνεύμα γειτονία, με, καλό, με πνεύμα καλής γειτονία, και λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή από τις ε, ενδιαφερόμενε χώρες. Στο αρχικό κείμενο του ψηφίσματος απευθύναμε και έκκληση στην ύπατη εκπρόσωπο κυρία Άστον και στον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Διεύρυνση να δραστηριοποιηθούν ακόμη περισσότερο υπέρ της επιλύσεως του προβλήματος που ακριβώς αυτό είναι το, εκεί το πρόβλημα, εκείνο το τείχος του Βερολίνου των εισαγωγικών που μπλοκάρει την πορεία της Μακεδονίας εδώ και 6 χρόνια. Αυτό είναι βεβαίως προς το συμφέρον της περιοχής, προς το συμφέρον της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα αρκεστώ σε αυτά, θα παρακολουθήσω προσεκτικά την συζήτηση θα ακούσω τα σχόλιά σας. Και ελπίζω να μπορέσουμε το ίδιο αποτελεσματικά και ευχάριστα να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Η κυρία Γιαννάκου παρακαλώ. Η κυρία Γιαννάκου. Α, ο κύριος Κούκαν πρώτα, ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή για την εργασία του Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες και εκφράζω την ελπίδα η Επιτροπή Εξωτερικών να εγκρίνει εν τέλει μια καλή ισορροπημένη έκθεση. Χρειάζεται η χώρα αυτή ενθάρρυνση στην πορεία της διότι έχει ανασταλεί η πορεία της για πολύ καιρό και αν συνεχιστεί αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω απογοητεύσεις και εντάσεις στη χώρα. Η λύση θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή ατζέντα. Χαίρομαι που η έκθεση ζητεί από το Συμβούλιο να επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Απηχεί η έκθεση ορισμένες από τις ανησυχίε που σημειώθηκαν στην τελευταία περίοδο. Επίση, οι επικείμενε εκλογέ θα είναι και καλύτερη ε, λύση για την χώρα. Αναμένουμε επίσης προόδους σε θέματα δημόσιας δικαιοσύνης, δικαιοσύνης και αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ελπίζω επίσης το μέγα θέμα να λυθεί σύντομα. Βρήκαμε κοινό έδαφος και με άλλες πολιτικές ομάδες για συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως εγώ υπεσχέθη να ζητήσω ορισμένες προσαρμογές στις συμβαστικές τροπολογίες. Ιδίω για την 2 κατά τμήματα ψηφοφορία για τα θέματα των ε, μειονοτήτων. Το ίδιο συμβαστική 7 για τις μακεδονικές αρχές να διαγραφεί η λέξη μακεδονικές και να λέει μόνο αρχές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Η κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι η έκθεση του κυρίου Τάλερ ε, κρατά σε μεγάλο βαθμό κάποιες ισορροπίες περιέχει όμως ορισμένα στοιχεία για να μην επαναλάβω και την επιχειρηματολογία ε, την οποία ανέπτυξα και άλλωστε αυτά θα τα ε, πει ο δικός μας shadow rapporteur ο κύριος Κούκαν ε, περιέχει ορισμένα σημεία και πάλι θα πρέπει κατά οριζόντιο τρόπο να φύγει η έννοια Ethnic Macedonia και Μασεντόνια σε όλη την έκθεση και βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί διότι ζητείται άμεση ε, έναρξη διαπραγματεύσεως αυτό που σημειώθηκε και πριν ότι η διαπραγμάτευση ε, βεβαίως αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά η απόφαση ανήκει στο Συμβούλιο. Η απόφαση για την ένταξη νέων χωρών ανήκει στις κυβερνήσεις και είναι αποκλειστικό δικαίωμά τους σε κάθε περίπτωση και είναι αποκλειστικό δικαίωμα και της κάθε μιας κυβέρνησης χωριστά. Και θέλω να σας επαναλάβω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα δεχθεί έναρξη διαπραγμάτευσης χωρίς λύση του θέματος. Ισχυρίζονται ορισμένοι ότι η Ελλάδα παρεβίασε την ενδιάμεση συμφωνία. Αλλά την παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας την έκανε η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η οποία ποτέ δεν χρησιμοποίησε το προσωρινό όνομα. Επομένως αυτό το θέμα θα πάει βέβαια ε, στη Χάγη και θα απαντηθεί εκεί, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσο περισσότερο πιέζεται η ελληνική πλευρά αδίκως για την υπόθεση αυτή, τόσο έξω θα μένει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και εάν αυτό το συνειδητοποιήσουμε θα πρέπει να στρέψουμε τις πιέσεις και τα βλέμματά μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι πρέπει να σας πω ότι ε, πριν από λίγο καιρό ε, η, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επεσκέφθη το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ρώτησε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς πάει το πράγμα και απήντησε ότι ο κύριος Νίμιτς έκανε μια πρόταση συγκεκριμένη, η Ελλάδα τη δέχθηκε και η άλλη πλευρά δεν είχε απαντήσει. Νομίζω λοιπόν πως η έκθεση του κυρίου Τάλερ αντί να ζητάει άμεση ε, έναρξη διαπραγματεύσεων καλό είναι να ζητήσει από την κυβέρνηση ε, της ε, ΦΥΡΟΜ να κάνει αυτά που πρέπει διότι διαφορετικά δεν υπάρχει καμία ελπίδα να, γίνουν, να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Κοπά και ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Ζόραν Τάλερ για την πληρέστατη και πολύ έντιμη έκθεση την οποία κατέθεσε ε, συζήτηση στην Επιτροπή μας ε, πραγματικά αντανακλά σε όλα τα επίπεδα την κατάσταση ε, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα ήθελα ε, απλώς να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κύριου Κούκαν επειδή ο όρος macedonian authorities αφορά το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης σήμερα στα ηνωμένα έθνη να τηρηθεί η πρακτική των προηγούμενων χρόνων και όπου αναφέρεται χαρακτηρισμός που αφορά τη χώρα να χρησιμοποιηθεί authorities of the state ή authorities of former ε, Yugoslav Republic of Macedonia. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πόσελτ. Πολύ σύντομα, διότι δεν θέλω να υπάρξουν παρανοήσεις. Γνωρίζουμε την πραγματικότητα και οφείλουμε να τη λάβουμε υπόψη. Ωστόσο, Θέλω να πω το εξή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διεξάγεται συζήτηση περί της ονομασίας. Η χώρα αυτή λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία κανένας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της ονομασίας αυτής. Μία και μόνη χώρα έχει πρόβλημα με την ονομασία αυτή εξού και το θέμα αυτό είναι διμερές. Επειδή λοιπόν η κατάσταση, η θεσμική κατάσταση είναι τέτοια όπως εξήγησε η κυρία Γιαννάκου, έχει γίνει και δικό μας το πρόβλημα. Λέω όμως σαφώς ότι δεν θέλουμε το πρόβλημα αυτό να επιβαρύνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνώ επίσης και με τα πλείονα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές και θα ξαναπώ, έστω και αν σας φανεί σαν ψευδέστηση, ότι θα πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως από την επίλυση μη διμερών θεμάτων, τα οποία διμερή θέματα μπορούν να επιληθούν στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν απαραίτητο να επιληθούν πρώτη ενάρξεως των διαπραγματεύσεων. Μέχρι την κύρωση της Συμφωνίας Εντάξεως μπορεί να λυθεί, όπως έγινε και στην περίπτωση Σλοβενίας-Κροατίας εγώ είμαι εισηγητής της ομάδας μας για θέματα Κροατίας. Δεν υπήρχε εκεί η προϋπόθεση να επιληθούν όλα τα προβλήματα μεταξύ Σλοβανίας, Σλοβενίας και Κροατίας πρώτης ενάρξης των διαπραγματεύσεων. Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, λύθηκε το πρόβλημα και ούτως ή άλλως ήταν αρκετά δύσκολο και έτσι. Κύριε Τάλερ παρακαλώ, στα σχόλια του συναδέλφου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρατηρήσεις και τις θέσεις που αναπτύξατε. Η ιστορία της Δημοκρατίας Μακεδονίας είναι καλά γνωστή σε όλες και όλους μας που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στην αίθουσα. Ούτε μπορούμε να επινοήσουμε κάτι τι το νέο. Υπάρχουν στο ψήφισμα κάποιες προτάσεις σχετικά. Προσωπικά ελπίζω ε, είπατε εκπροσωπή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, να φανούν ακόμα πιο δραστήριοι σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τις δύο πλευρές να ψάξουν και να βρουν μια λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για πάντα. Το αδιέξοδο, η κατάσταση αυτή όπου δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι ουδέτερη, είναι αρνητική. δεν είναι μια διαδικασία που επιτρέπει να μην τα πράγματα ως είναι, διότι προκαλεί πολλή απογοήτευση και ενδεχομένως να είναι απαρχή αρνητικών εξελίξεων, όχι μόνο στην ίδια τη χώρα αυτή, αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια. Θα ζητήσω λοιπόν και πάλι υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Αυτή είναι και η πρόταση που κάνει το ίδιο το ψήφισμα. αναμένοντας την ψηφοφορία του απογεύματος και τις ε, τελικές μας αποφάσεις της επόμενης Ολομέλειας. Σας ευχαριστώ. Έτσι μας δίνεται μια ιδέα για το πώς να προχωρήσουμε παραπέρα και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή στην έκθεση του κυρίου Προβέρας για τα μεταναστευτικά ρεύματα που προκύπτουν από την αστάθεια. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο εισηγητή να λάβει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άτυπα, όχι επίσημα εν πάση περιπτώσει, αλλά να συγχαρώ ειλικρινά τους σκιώδεις, οι οποίοι εργάστηκαν εξαιρετικά με πολύτιμες υποδείξεις οι οποίες ελήφθησαν υπόψη και εντάχθηκαν στην έκθεση. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους Κρέτσου και Κέλλερ, ε, εξ ονόματος της Ντέβε και Λίμπε, από την Ντέβε και Λίμπε, και τη γραμματεία η οποία μας βοήθησε πραγματικά. Τέλος, να ευχαριστήσω τους συντονιστές ε, διότι με την εμπιστοσύνη τους μου με άφησαν να εργαστώ επί μιας έκθεσης στην οποία πιστεύω ειλικρινά εδώ και πολύ καιρό. Δεν θα επαναλάβω τους λόγους που με οδήγησαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης και στις υποδείξεις και τα χαρακτηριστικά της. Θα ήθελα να υποστηρίξω στο ότι εν λόγω έκθεση είναι επίκαιρη με βάση την ε, κατάσταση στις χώρες ε, Μασρέγ και Μαγκρέμπ. Έχουμε 168 τροπολογίες και φτάσαμε σε 9 τροπολογίες συμβιβασμού. Τρεις θα είναι προφορικές. και θα τη συζητήσουν οι υπογράφοντες, οι συντάκτες. Ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι η κατάσταση της Λιβύης ε, με την αναστολή διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λιβύης, της Συμφωνίας Πλαισίου, για σαφείς λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Για την ε, μεγάλη αναταραχή σε αυτή τη χώρα. Ελπίζουμε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις όταν συσταθεί μια κυβέρνηση που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των μεταναστευτικών ροών που προέρχονται από την νότια όχθη της Μεσογείου μαζί με τις μεταναστευτικές ροές εξανατολών. Έχουν ενταχθεί και τροπολογίες συμβιβασμού που αναφέρονται σε ορισμένες ευάλωτες ομάδες, εθνικές ομάδες και έχουν ενταχθεί και ορισμένες τροπολογίες που αφορούν και τις φυσικές καταστροφές ως αίτιο μεταναστευτικών ροών. Κλιματικές αλλαγές, αστάθειες και ούτω καθεξής. Γνωρίζετε το περιεχόμενο της έκθεσης στις μεγάλες ε, ευρείες αδρές γραμμές και με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μοντάλτο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Προβέρα διότι μπόρεσε να, οδηγήσει, να καθοδηγήσει τους σκιώδεις κατά τρόπον ώστε όποιος διαβάσει αυτή την έκθεση να αναγνωρίσει το γεγονός ότι είναι μία ισορροπημένη έκθεση. Η μετανάστευση είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα αρκεί να κοιτάξουμε πώς το αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης ή τα πολιτικά κόμματα. για το τι περιλαμβάνει μετανάστευση, πώς, πώς ορίζεται, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις ενδοκινοτικά δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν σε μία έκθεση η οποία εστιάζει την προσοχή στην εξωτερική μας πολιτική για την αντιμετώπιση αυτών των μεταναστευτικών φαινομένων. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ορισμός αστάθεια είναι ιδιαίτερα εύρης και αυτή είναι η λέξη κλειδί που αφορά αυτή την έκθεση. Πρόκειται για μια την ευρύτερη δυνατή έννοια έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση με βάση τις υποδείξεις των ε, διαφόρων εισηγητών για να μιλήσουμε για ανθρώπινα φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, αποψήλωση, κλιματικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Μιλάμε δηλαδή και για ανθρωπογενή ε, φαινόμενα όπως και καταστάσεις πολιτικής κρίσης. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους άλλους ε, σκιώδεις, διότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Έχω υποβάλει μία τροπολογία η οποία ε, ξεπεράστηκε από τα γεγονότα και ίσως πρέπει εγώ ίδιος να την καταψηφίσω διότι ε, ξεπεράστηκε από τα γεγονότα. Για άλλη μια φορά θα ήθελα εν συμπεράσματι να πω ότι η έκθεση αυτή θα λάβει τελική μορφή, βρίσκεται εν εξελίξη και στην τελική της μορφή θα πρέπει να αποφανθεί για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο βρίσκεται ε, σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης. Μπενάρα Πάτου. Λόπες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Προβέρα για την έκθεση για τις μεταναστευτικές ροές, διότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Πρέπει να συζητηθεί εδώ στην ΑΦΕΤ, συνήθως αφορά τη ΛΥΜΠΕ. Και μας απασχολούν θέματα ασφάλειας. Πολλές φορές η οπτική μας γωνία είναι διαφορετική. Εδώ μιλάμε για τα διεθνή φαινόμενα που είναι απότοκα αυτό των μεταναστευτικών ροών και πώς θα συνεργαστούμε με τις χώρες διαμετακόμισης αλλά και καταγωγής. Η οπτική μας γωνία είναι πολύ σωστή και μέσα στα πλαίσια της ε, διεθνούς μας ε, πολιτικής δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το θέμα ασφάλειας. Είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας γενικότερα, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε αυτές τις ροές, γιατί τις θεωρούσαμε πάντα απειλή. Δεν τις είδαμε υπό διαφορετική οπτική και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και αυτές τις ε, ε, μεταναστευτικές τάσεις και το πώς επιδρούν επί του μέλλοντός μας. Θα πρέπει να έχουμε απτά στοιχεία, διότι πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ προσφύγων, ετούντων άσυλο, μέσα στα πλαίσια της σύμβασης της Γενέβης ή είναι πρόσφυγες διότι ζητούν προσωρινή προστασία διότι δεν μπορούν να ενταχθούν στη σύμβαση της Γενέβης γιατί ζητούν επικουρική βοήθεια ή γιατί μιλάμε για μεταναστευτικές ροές μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης κινητικότητας για αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. και γιατί αποζητούν οι μετανάστες ε, ε, εργασία μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει πιο λεπτομερής ανάλυση για να γνωρίσουμε καλύτερα τα γεγονότα, να έχουμε απτά στοιχεία και να μπορούμε να εντάξουμε αυτά τα στοιχεία στις διεθνείς μας σχέσεις, δηλαδή να υπάρχει ένα συσχετισμός με άλλες χώρες υπό μια άλλη οπτική θεώρηση μέσα στα πλαίσια της ε, ΛΥΜΠΕ, όπου είμαι πλήρες μέλος και όπου θεωρείται η μετανάστευση ως απειλή. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την έκθεση και ελπίζω στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές ως έχουν και να διαχωρίζουμε τα διάφορα επιμέρους φαινόμενα. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δημιουργούνται ε, δύσκολες καταστάσεις για τις χώρες καταγωγής ή τις χώρες διαμετακόμισης. Ο κύριος Πρωτασέβης. Θα μιλήσω πολωνικά, συνάδελφοι, με την άδειά σας, εφόσον υπάρχει διερμηνία. Θα... Ή ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Είχαμε επικοδομητικές ε, διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθαμε σε επαφή με τους διάφορους εκπροσώπους πολιτικών ομάδων και νομίζω ότι οι θέσεις μας αντικατοπτρίζονται πολύ καλά. Μιλώ εξ ονόματος του ΕΛΚ, αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός αφορά και πολιτικά γεγονότα. Γεγονότα τα οποία... Ε, επισυνέβησαν στο μεταξύ από την ε, στιγμή της σύνταξης μέχρι τη σημερινή στιγμή που συζητάμε την έκθεση αυτή. Βλέπουμε τα πολιτικά γεγονότα, τα δραματικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Λιβύη, που θα έχουν επίπτωση στην τελική σύνταξη της έκθεσης ως προς τις μεταναστευτικές ροές. Διότι οι μεταναστευτικές ε, ροές είναι απότοκες των κλειδονισμών σε αυτή την περιοχή της Βορείου Αφρικής και θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή γιατί μπόρεσε να προσαρμόσει την έκθεσή του και να ανταποκριθεί στα πραγματικά γεγονότα. Χαίρομαι, διότι πολλές ιδέες ε, εντάσσονται σε αυτή την έκθεση και θα ήθελα να στραφώ στην παράγραφο 4 και στο τι αναφέρεται εκεί. Μιλάμε για την αιρεσιμότητα. Όταν διαβάσουμε την παράγραφο 4 βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ερεσιμότητα, δηλαδή όροι που να διέπουν την ε, δική μας βοήθεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει χρηματοοικονομική βοήθεια μέχρι ότου είμαστε απόλυτα σίγουροι, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αφρικανικών χώρων, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων πολιτικών και οικονομικών. Και οι κλειδονισμοί που γνωρίζουμε ε, αφορά έλλειψη βοήθειας από εμάς στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε δικτάτορες και ούτε καν τις κυβερνήσεις αλλά τον ε, μέσο πολίτη γιατί εάν οι άνθρωποι ζουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, τότε δεν θα διακινδυνεύουν να έρχονται στην Ευρώπη ως παράνομοι μετανάστες. Προέρχομαι από μια χώρα που εντάχθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το βορρά, από τα βόρειο-ανατολικά σύνορα που έχουμε περιορισμένη πείρα σε σχέση με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία ή την ε, Μάλτα. Η πείρα μας στην Πολωνία είναι πολύ περιορισμένη, αλλά αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει. Και ο εισηγητής δίνει πολλές συστάσεις για το πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε με την παράνομη μετανάστευση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιμερίσουμε αυτό το άχθος, αυτό το φόρτο και θα πρέπει να αναφερθούμε στην πάγια αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πρόκειται για θεμελιώδη αξία αυτής της έκθεσης. Και τέλος, ε, Πρόεδρε, στο, στη Συμφωνία συμβιβασμού, στις τροπολογίες συμβιβασμού μιλάμε για συνεπείς λύσεις ως προς τη μετανάστευση και την νόμιμη. Θα χρειαστούμε μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αποτελεί καινοτόμο στοιχείο, αλλά υπάρχουν πολιτικές από ΙΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και θα πρέπει εμείς να έχουμε τη δική μας μεταναστευτική πολιτική. Μια συνεκτική πολιτική σε σχέση με τη μετανάστευση από άλλες χώρες. Διαφορετικά θα έχουμε τους χειρότερους δυνατούς μετανάστες και αυτό το λέω μέσα σε εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Προβέρα. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως το θέμα με το οποίο ασχολείται είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος. Και θα συμφωνήσω με την άποψη ότι ίσως θα έπρεπε να δούμε το θέμα όχι μόνο από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας αλλά από πλευράς οικονομικών επιπτώσεων, κοινωνικών επιπτώσεων και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και να το δούμε σοβαρότατα και όχι μόνο στη θεωρητική του βάση. Διότι φοβάμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις συστάσεις του κυρίου Προβέρα και άλλων εισηγητών της Λίμπη από ό,τι άκουσα από την κυρία, βλέπουμε επιφανειακά το θέμα. Το θέμα φοβούμε ότι γίνεται ουσιαστικότερο και θα είναι το μέγα πρόβλημα της προσεχούς 20 κυρίως για την Ευρώπη. Από στατιστικές που είδα, 7.400.000 νέοι ηλικίας από 19 έως 27 ετών ζητούν εργασία στην Ευρώπη. Μας λείπουν περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή όμως παρότι λείπουν τόσες θέσεις εργασίας έχουμε τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα. Από την άλλη πλευρά γυράσκει ο πληθυσμός της Ευρώπης. Το 2030 υπολογίζεται ότι η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων θα είναι 430 από αυτόχθονες Ευρωπαίους. Την ίδια χρονική περίοδο από στατιστικές που βλέπω και με τρομάζουν στην κυριολεξία κύριε Πρόεδρε βλέπουμε ότι ε, Ισλαμικοί πληθυσμοί που σήμερα ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο 600 εκατομμύρια το 2030 θα είναι 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια. Δηλαδή μια καινούρια Ευρώπη και κάτι παραπάνω, μια Ευρώπη πλάς γεννιέται στον πλανήτη. Είναι φυσικό λοιπόν όπου αφήνονται κενά να μπαίνει ε, σαν νερό, σαν, ε, σαν ποταμός κάποιο άλλο στοιχείο, διότι στη φύση πάντα υπάρχουν ισορροπίες που πρέπει να καλυφθούν, που να ε, μπορέσει να το καλύψει. Αυτό μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι θα έχουμε ανατροπές στην Ευρώπη, τόσο από πλευράς οικονομικής, όσο και από πλευράς κουλτούρας και εν πάση περιπτώσει και ασφάλειας, διότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί πώς θα αντιμετωπιστούν στην Ευρώπη με τις ροές οι οποίες υπάρχουν από πλευρά υγείας παραδείγματος χάρη. Έχουμε τις υποδομές να τους προσφέρουμε την κατάλληλη υγεία. Ε, έχω το παράδειγμα στην πατρίδα μου στην Ελλάδα όπου ιδιαίτερα στα νοσοκομεία παιδών εμφανίζονται οι πληθυσμοί των ε, ασθενών ε, λάθρομεταναστών κυρίως στο 90% των πελατών και έχουμε ένα 10% Ελλήνων ασθενών να πάνε να νοσηλευτούν. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει επέλθει μια τεράστια ανατροπή. Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ανατροπή οικονομική. Διότι όλη αυτή η κατάσταση έχει ένα κόστος λειτουργίας νοσοκομείων, λειτουργίας ε, φαρμακευτικής περιθάλψεως κτλ, κτλ. Το οποίο αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να το αντιμετωπίσουν και πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα λοιπόν εν κατακλείδη για να μην σας κουράζω, διότι αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας έχουμε το θέμα αυτό, το έχουμε πάρει στα σοβαρά, να μην μείνουμε στη θεωρία του θέματος. Να κάνουμε κοινέ ενέργειες και συντονισμένες πρακτικές να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα το λύσουμε, αλλά απλώς θα το αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Κύριε Προβέρα, αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Με μεγάλη ειλικρίνεια θα πω ότι οι συνάδελφοί μου τόνισαν θέματα που και εγώ θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά και που ίσως δεν έχουν περιληφθεί όλα στην έκθεση, αλλά αυτό έχει σχέση και με τα θέματα αρμοδιοτήτων. Εμείς είμαστε Επιτροπή Εξωτερικών και δεν θα πρέπει να αναμειχθούμε σε αρμοδιότητες άλλων, ε, άλλων επιτροπών. Θα αρχίσω πρώτα από τον κύριο Μοντάλντο, που αναφέρθηκε στις βάσεις της εκθέσεως. Γίνεται δηλαδή η προσπάθεια να τεθεί το θέμα στις ιστορικές του διαστάσεις αλλά και με τρόπο διακομματικό. Βέβαια, συνέβαλαν με τις θέσεις τους διάφορα πολιτικά κόμματα. Πάντως αυτή είναι η δική μου προσπάθεια να κάνω μια υπερκομματική θεώρηση. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Λόπες επίσης, επίσης και άλλωστε η δική μας προσέγγιση εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών είναι διαφορετική από ό,τι άλλων επιτροπών. Προσπαθούμε να φωτίσουμε το πρόβλημα από όλες τις πλευρές και πέραν των ειδικών συνθήκων του παρόντος. Όπως είπα, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε από πολλές πλευρές. Και εάν κάποια στιγμή είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να λειτουργήσει προληπτικά σε χώρες με ασθενείς ιστούς, τότε θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και ως Ευρωκοινοβούλιο να, έρθουμε, να φέρουμε σε ισορροπίες τις δράσεις μας και με άλλες χώρες και όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Κίνα και τη Ρωσία επικαλύψεις και περιττός ανταγωνισμός θα πρέπει να αποφευθούν, διότι αλλιώς δεν θα είναι αποτελεσματικές οι δράσεις που θα αναλάβουμε. Η κυρία Λόπες έχει επίσης δίκιο όταν λέει ότι τη μετανάστευση δεν πρέπει να την θεωρήσουμε μόνο ως απειλή, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ μονομερές. Η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει και πόρο και για τις χώρες αποστολής μεταναστών και για τις χώρες υποδοχής μεταναστών αλλά πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική με ξεκάθαρους κανόνες για να βασιστεί σε αυτούς μια συνεργασία για καλύτερα αποτελέσματα. Για σας κύριε Πρωτασίεβιτς. Όλοι παρακολουθούμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και νομίζω και γι' αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος της Επιτροπής Εξωτερικών που πρέπει να ρίξει το βάρος της και σε μια προσπάθεια πρόληψης των προβλημάτων αυτών που έχουν κάποια σχέση με προβλήματα υποδομών και δομών. Είναι η Επιτροπή μας εκείνη η οποία μπορεί να αντιδράσει στις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο για το άρθρο 4, για την ερεσιμότητα. Παράγραφος 4. Ερεσιμότητα. Ε, δεν, είναι, δεν σημαίνει ε, ε, ότι εκβιάζουμε ή επιβάλλουμε όρους με την ερεσιμότητα ή είναι κάτι το οποίο είναι απότοκο των εθνικών μας συμφερόντων. Ερεσιμότητα σημαίνει αποδοτική παρέμβαση για τους ανθρώπους. Εγώ παρακολουθώ την διεθνή συνεργασία εδώ και 20 χρόνια. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Οι περισσότεροι πόροι που καταβλήθηκαν από κράτη, μεμονωμένα κράτη ή από διεθνείς οργανισμούς ή υπεξαιρέθηκαν επί της ουσίας και οι άνθρωποι δεν έλαβαν σχεδόν τίποτα. Άρα αιρεσιμότητα σημαίνει αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και αυτό αφορά τις συνθήκες in situ και με την καλύτερη δυνατή θέληση δεν μπορούν να πραγματοθούν, να υλοποιηθούν σχέδια εάν δεν υπάρχει προσβασιμότητα ή αν δεν υπάρχουν οδικές αρτηρίες, για να πω κάτι το, το πολύ αυτονόητο. Δύο λεπτά ακόμα, Πρόεδρε, αλλά το θέμα είναι, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αιρεσιμότητα αφορά και τη σταθεροποίηση ορισμένων ε, καταστάσεων. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε χώρες χωρίς να απαιτούμε ε, μία κατάσταση, μία πολιτική κατάσταση υπέρ της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε δικτατορικές χώρες ή ψευδοδημοκρατικές χώρες, διότι σε αυτή την περίπτωση ε, ενισχύουμε τη θέση του κυβερνώντα κατά του λαού. Αυτό είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τέλος, σε σχέση με το συνάδελφο Προτασχέβης, θα ήθελα να πω ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική βεβαίως προβλέπει, προβλέπει τις ε, καταστάσεις παρανομίας, διότι είναι ένα δεδομένο. Αλλά μία πολιτική μετανάστευση θα πρέπει να είναι συνεπής ε, με αυτά που είπαμε πριν προς τον κύριο Σαλαβράκο. Ο κύριος Σαλαβράκος έθιξε ένα ζήτημα το οποίο είναι ύψης της σημασίας, ιδιαίτερα για τις χώρες του τρίτου κόσμου. Τι ζητούν οι περισσότεροι, πολλές, αρκετές χώρες, σε πάση περιπτώσει. Και από τη δική μας Ήπειρο, ακόμα. Τι ζητάμε από τη μετανάστευση. Πολλοί θέλουν οι, οι μετανάστες να είναι νέοι, να έχουν επαγγελματική κατάρτιση, να είναι καλλιεργημένοι, να έχουν προσόντα που να είναι χρήσιμα για τις κοινωνίες μας. Μα συνάδελφοι, αυτό οδηγεί στο brain drain. Δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε τους καλύτερους εγκεφάλους από αυτές τις χώρες που είναι χώρες αναπτυσσόμενες και τις καταδικάζουμε σε μια καθυστέρηση αναπτυξιακής πορείας με αυτή την απορρόφηση εγκεφάλων. Δηλαδή προβαίνουμε στην αποστράγγιση αυτών των χωρών. Υπάρχουν οικονομικά θέματα, κοινωνικής υφής, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για πολιτισμικές αξίες. Προσπάθησα να το δω το θέμα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά μπορούσα. Σας ευχαριστώ ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ε, Μουλτσουμέσκ, είπε ο κύριος Προβέρα στα ρουμανικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα και θα πρέπει να το γνωρίζετε. Τώρα συνεχίζουμε στο τελευταίο θέμα. Τη ημερήσια διάταξη για το πρωί. Απαλλαγή 2009. Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα 3, Επιτροπή. Στο σημείο 9. Α, να δώσω το λόγο στην κυρία Βερονίκη Τικάιζερ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για ένα θέμα το οποίο δεν παρουσιάζει τόσο ζωηρό ενδιαφέρον, δηλαδή το θέμα της απαλλαγής. Όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί θα δούμε κατά πόσο οι δαπάνες των θεσμικών οργάνων έτυχαν επαρκούς ρυθμού εκτέλεσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους μας, τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ε, τεχνικό αυτό εγχείρημα προετοιμάζεται από το ελεγκτικό με μια σειρά εκτιμήσεων, αξιολογήσεων και συστάσεων που βρίσκονται μεταξύ σελίδας 136 και 159 και πρόκειται και για ένα πολιτικό εγχείρημα διότι θέλουμε και εμείς να αποφανθούμε για το κατά πόσο αυτό ήταν το ζητούμενο. Μιλάμε για πέντε παραγράφους και για να κινηθώ εντάχει θα ήθελα να πω ότι συνιστώ την απαλλαγή με βάση την έκθεση του ελεγκτικού. Μία τώρα γενική σύσταση, μάλλον ένα σχόλιο, είναι ότι υπάρχει μείωση σφαλμάτων σε σχέση με τα παρελθόντα ότι υπάρχουν ε, λάθη εξ άντε και εξ post, αλλά γενικά η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Διαγράφεται μια θετική τάση και γι' αυτό το λόγο ε, προβάλλω και θετική άποψη, υπέρ δηλαδή της απαλλαγής. Όταν δούμε την έκθεση σε λεπτομέρεια του ελεγκτικού, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα. Όμως Ε, υπάρχουν σαφέστερες ε, θετικές τάσεις για το μέλλον. Δηλαδή γίνεται πολύ καλή χρήση των δεδομένων και αυτό θα το δούμε και μακροχρόνια. Υπάρχει ε, ένας αριθμός φαλμάτων για το έτος 2009 για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σφάλματα εκλογιμότητας ως προς την επιλεξιμότητας ως προς τις δημόσιες προμήθειες. Δέχομαι ε, τα δεδομένα του ελεγκτικού συνεδρίου που αναφέρεται τα σφάλματα πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό είναι προφανές. Όμως, για ορισμένα από αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να δεχτούμε μερικά από αυτά διότι οι καταστάσεις είναι ασταθείς, δεν μπορούν να οριοθετηθούν. Μιλάμε για το μέσο σταθερότητας, μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο και ούτω καθεξής. Άρα Εάν κινούμαστε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές, τότε μπορούμε να ανεχτούμε και ορισμένα ασφάλματα. Για τα υπόλοιπα, μπορώ να πω ότι κινούμαστε προς τη μηδενική ανοχή, μακροχρόνια, και οι διατάξεις είναι σωστές και η θέση της Επιτροπής ικανοποιητική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Λέζιν και Μακοβέι της Σκιώδης. Υπάρχουν πέντε τροπολογίες. Μπορώ να δεχτώ το, δηλαδή δέχομαι το σκεπτικό της κυρίας Λέζινγκ, αλλά δεν μπορώ να τις δεχτώ τελικά. Δεν μπορώ να δεχτώ τις δύο και τρία. Τις άλλες τροπολογίες μπορώ να τις δεχτώ. Της κυρίας Μακοβέη δηλαδή. Στην τροπολογία 2, η κυρία Σαμπίνε Λέζινγκ προβάλλει μία τροπολογία, υποβάλλει μία τροπολογία πολιτικής καθαρά χρειάς, που είναι ευπρόσδεκτη κάθε αυτή, αλλά η οποία τονίζει στο ότι ο, ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις κατευθυντήριε γραμμές ως προς την εξωτερική πολιτική και να είμαστε μια ειρηνική δύναμη και να δράσουμε ως μεσολαβητής ε, για την ειρηνική επίλυση ε, σειράξεων, το becomes. Μα μέχρι τώρα δεν ήμασταν, ε, ήμασταν φιλιρινικοί πάντα. Άρα το becomes δίνει λανθασμένη εντύπωση. Ποτέ δεν είχαμε ταχθεί υπέρ μιας ε, βίαιης λύσης. Είμαι υπέρ μιας Ευρώπης της άμυνας και στα πλαίσια του ε, διεθνούς δικαίου, όπως ε, συζητήθηκε στο Στρασβούργο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια στρατιωτική δράση αν εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή δεν λέμε ότι εμείς είμαστε φιλιρινιστές και οι άλλοι, το ΝΑΤΟ και άλλες δυνάμεις σας κάνουν, οι άλλοι οργανισμοί σας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αποκλείουμε εξαίρεση κάτι διαφορετικό για να μην προβάλλω μία προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας δεν θα τη δεχτώ τη 2 θα την απορρίψω τη 2 τώρα ως προς την τροπολογία 3 η κυρία Λέζινγκ προβαίνει σε μία διαγραφή το ότι δηλαδή δέχομαι ένα περιθώριο λάθους σε έκριθμες καταστάσεις όταν μιλάμε για ε, διεθνείς σειράξεις, ex δηλαδή δεν δέχομαι την αρχή λάθους, αλλά δέχομαι τα περιθώρια λάθους και θα ήθελα να παραμείνει το κείμενο ως έχει. Αυτά έχω να πω. Δεν είναι και πολλά, αλλά νομίζω ότι ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι χορηγούμε την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λόζενγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ντεκάιζερ η οποία με τόσο επισταμένα ασχολήθηκε με τις τροπολογίες μου. Λυπάμαι ασφαλώς που δεν συμφωνεί με την τροπολογία αυτή για την ειρηνική εξωτερική πολιτική γιατί στην αρχή μου είχε δοθεί η εντύπωση ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει. Αλλά τελικά δεν συμφώνησε. Αυτή την τροπολογία δεν πρόκειται να την ε, τροποποιήσω γιατί δεν ε, ανταποκρίνεται στα πιστεύω μου και δεν ανταποκρίνεται και στα πιστεύω της ομάδας μου αυτό που προτείνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κοιτάξω τα υπόλοιπα σημεία τα οποία θίξατε και στο τέλος, σε ό,τι αφορά την παράγραφο 4, σε περίπτωση που μιλάτε για ποσοστό σφαλμάτων και την ανοχή για το ποσοστό αυτό, ε, εξηγήσατε τι εννοείται, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή ε, δίνουμε μια λευκή επιταγή για τέτοιο ποσοστό σφαλμάτων. Δεν είναι δύσκολο θεωρώ στο GSP να χρησιμοποιήσουμε τα επιχειρήματα που αναφέρατε και η επιχειρηματολογία είναι πολύ γενική. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζήτησα να διαγραφεί, να διαγραφεί η παράγραφος 4 και θα, δεν θα αποσύρω την τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Ντεκάιζερ. Madame Kaiser, would you like to react? Όχι. Σέβομαι τη θέση της ε, κυρίας Λέζινγκ. Απλώς ε, εγώ μίλησα για έκτακτες καταστάσεις καθόλου έκτακτες καταστάσεις. Καταλαβαίνω όμως και τη δική, σας, τη δική της θέση. Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα για την έκθεση αυτή. Και άρα θεωρώ ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση και θα τα πούμε το απόγευμα στις 3. Στην ίδια αίθουσα. Σας ευχαριστώ. <laughs>